Ja, guten Tag. Wir Ξαναρχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και στην ε, ημερίδα εργασίας για την καταπολέμηση της, ε, του ευτροφισμού στην Βαλτική με τον κύριο Σαουάρμα, εισηγητή. Σας καλωσορίζω κύριε Βέρμα, κύριε Λουρουά, κύριε Κόρμπινεν, Τόρινσεν, Τελένσκι. Περιμένουμε βεβαίως να μας ενημερώσετε για την κατάσταση και βέβαια σε συνάφεια με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ξεκινούμε με τον κύριο Σαβουάρμα που παίρνει το λόγο σύγητης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, και τους καλεσμένους μας που είναι παρόντες. Ε, και ευχαριστώ ιδιαίτερως τους εμπειρογνώμονές μας. Είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας σε αυτό το σημαντικό σεμινάριο, εργαστήριο. Και μακάρι και περισσότεροι ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Γιατί ενημερώσαμε και στην επίσημη ιστοσελίδα μας για την εξαγωγή αυτού του σεμιναρίου. Η Βαλτική θάλασσα είναι από τις πιο μολυσμένες, ρυπασμένες θάλασσες ε, του κόσμου και ο ευτροφισμός των οικοσυστημάτων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της περιοχής. Και δεδομένων των αυτών αποτελεσμάτων στο περιβάλλον, ο ευτροφισμός επηρεάζει ε, και 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή ε, της Βαλτικής. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας ε, και με έγκριτους ε, εμπειρογνώμονες ε, θα κατατοπιστούμε περισσότερο. Πριν δύο χρόνια, το 2016, υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού το έγγραφο εργασία για μια ειδική έκθεση που έγινε από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο με τίτλο «Η καταπολέμηση του ευτροφισμού στη Βαλτική θάλασσα». Χρειάζεται περισσότερη και πιο αποτελεσματική δράση. Ε, ένα από τα σημαντικότερα πορίσματα της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2016 ήταν ότι παρά τη σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση του ευτροφισμού της Βαλτικής θάλασσας είναι δυστυχώς πολύ περιορισμένη. Στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη, στα σχέδια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων στις ε, παραθαλάσσιες περιοχές ήταν 14,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 44 εκατομμύρια ευρώ στηρίζοντας παρόμοια συναφή σχέδια στη Λευκορωσία και Ρωσία. Σε αντάλλαγμα για τα κονδύλια που δόθηκαν στον αγώνα για την καταπολέμηση του ευτροφισμού ε, τα αποτέλεσματα ήταν μάλλον πένιχρα. Κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη πιο αποτελεσματικής προσέγγισης ε, και μεγαλύτερης ε, αξιοποίηση των κονδύλιων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και συγκεντρώσαμε πυρογνώμονες με βρυφάσμα γνώσεων για να καλύψουμε ολόκληρη την κατάσταση στη Βαλτική και χωρίσαμε σε τρεις ε, θεματικές οντότητες στην ε, σημερινή μας ακρόαση. Θα μιλήσουμε πρώτα για την κατάσταση στη Βαλτική γενικώ, ε, για τη συμμετοχή των ερευνητών και τα πορίσματά του για τον ευτροφισμό και το τρίτο τμήμα θα αφορά τις διάφορες πολιτικές χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του ευτροφισμού. Μετά από κάθε θεματική ενότητα, μετά από κάθε πάνελ θα προβλέψουμε και ένα χρόνο για συζήτηση, για ερωταπαντήσεις και εκεί θα καλέσω τους συναδέλφους ε, να λάβουν μέρος στη συζήτηση για την αξιοποίηση των κοινωτικών κονδυλίων προκειμένου να καταπολεμηθεί ο ευτροφισμός, αυτή η μάστιγα της Βαλτικής. Και μάλιστα θα ήθελα να μην επικεντρωθούμε μόνο σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που επίσης ε, βρέχονται από τη Βαλτική και πώς θα συμπεριλάβουμε στην προοπτική μας και αυτές. Σας ευχαριστούμε. Όντως πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Το θέμα πρώτος ομιλικής μας είναι ο κύριος, η κυρία Βιβινίμενμα από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς απόγευμα. Και με χαρά θα σας παρουσιάσω τον δημοσιονομικό έλεγχο επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στις αρχές του 2016 κατά πολέμηση του ευτροφισμού στη Βαλτική είναι ο τίτλος. Κύριο Συμπέρασμα, χρειάζεται περισσότερη και πιο αποτελεσματική δράση. Ο ευτροφισμός λοιπόν τι είναι, προξενείται από υπερβολική ε, παρίσφρηση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, που μπορεί να έχουν και ε, τοξικές συνέπειες. Περιορίζει ο ευτροφισμός τη βιοπικιλότητα, περιορίζει τα ε, αποθέματα, την ανανέωση της θάλασσας. 95% λοιπόν της ε, Βαλτικής επηρεάζεται, παρουσιάζει φαινόμενα ευτροφισμού, ακόμη και αν ε, μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς. Υπάρχουν ε, δύο τύποι ρήπανσης αποθρεπτικές, καταρχάς η διάχυτη που προέρχεται από τη γεωργία και η ε, ρήπανση η σημειακή. Με κύριο αίτιο τα λίματα. Και αυτό αναφέρουμε και στην ε, έκθεσή μας. Επικριτικά λοιπόν τη γεωργία με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, Λετωνία, την Πολωνία και τη Φινλανδία και τα λίματα για τη Λετωνία και την Πολωνία. Και βεβαίως αντίστοιχα εξετάζουμε και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι οδηγίες που έχουν να κάνουν με τις θρεπτικές ουσίες, η μία που έχει να κάνει με τα νητρικά και τα αστικά λίματα ε, έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα όρια, ορίζουν συγκεκριμένα τα όρια για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόκειται ωστόσο για οδηγίες οι οποίες δεν έχουν επαρκέ αποτελέσματα όμως για τη Βαλτική, γιατί είναι ε, μια θαλάσσια ζώνη βαλτική ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Και έτσι έχουν ε, προταθεί ιδιαίτερες προδιαγραφές πέραν των ευρωπαϊκών με τη, συνθήκη, με τη σύμβαση του Ελσίνκη και αυτό βέβαια το υιοθετούν οι χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική συμπεριλαμβανομένες και της Ρωσίας. Οι δύο οδηγίες της 21ης, ε, του 21ου αιώνα έχουν μια προσέγγιση διαφορετική από τις προηγούμενες. θεωρούν ως σημείο κίνησης ένα καλό επίπεδο περιβαλλοντικό, δηλαδή για να επιτευχθεί το καλό περιβαλλοντικό επίπεδο πρέπει να αναλυφθεί κάθε προσήκον μέτρο και βεβαίως το επιπλέον κόστο, η διαχείριση των ε, κοιτών των ποταμών με την οδηγία για τα ύδατα ε, έχει όρους ε, ικανούς να περιορίσουν το πρόβλημα στη Βαλτική στην ελεκτική μας δραστηριότητα. Εξετάσαμε κυρίως αν ήταν αποτελεσματικές οι δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να κράτη-μέλη να περιορίσουν την παρουσία των ρηπογόνων ουσιών ε, και των θρεπτικών αυτών στη Βαλτική. Η απάντηση είναι μόνο περιορισμένη πρόοδος, έχει σημειωθεί, για τη γεωργία. Ήταν πλημελής ο προσδιορισμός των ε, ευάλωτων σε μητρικά ζωνών Επίσης, προγράμματα δράσεων σχετικά με τα νητρικά δεν είναι αρκετά αυστηρά από ό,τι διαπιστώνουμε. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στοχεύει επαρκώς σε μέτρα ανάπτυξη πέθρου για τις ε, ε, ζώνες που θα είχαν προς τώρα ανάγκη. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση, ιδιαίτερη στόχευση για τις ζώνες που παρουσιάζουν προς τώρα προβλήματα. Αλλά για να σας δώσω και κάποια καλά νέα, βλέπουμε βελτιώσει σε σχέση ε, με την νέα περίοδο 2014-2020. Στη συλλογή και επεξεργασία αστικών κλιμάτων. Διαπιστώνουμε ότι μόνο δύο έχουν πλήρω συμμορφωθεί με τη σχετική οδηγία, τη στιγμή τουλάχιστον ε, του ελέγχου. Η Πολωνία, παραδείγματι, παρά τι τεράστιε επενδύσει με συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ χαμηλή συμμόρφωση. Επίσης η αξιολόγηση της υλοποίησης των οδηγίων, της οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχωρεί με καθυστερήσεις, αλλά και πάλι έχουμε ένα καλό νέο, ότι δηλαδή οι μονάδες κατεργασίας λιμάτων που εξετάσαμε στην Λετωνία και την Πολωνία ε, έχουν ε, ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, χωρίς όμως εγγυήσεις οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς ορισμένες από αυτές είναι ε, υπερμεγέθης. Για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία τώρα τους γείτονες, πάλι βρίσκονται στην ίδια ζώνη της Βαλτικής, στη ζώνη των λεκανών απορροής. Έχουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της ε, βόρειας ε, γειτονίας με έργα αποτελεσματικά γιατί έχουμε να κάνουμε λίγο πολύ με όρημα φρούτα, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να περιοριστεί η αναλογία θρεπτικών σε σχέση με το κόστος σε ευρώ. Όπως είπα, ωστόσο ήταν περιορισμένη η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις επενδύσεις. Καλό νέο είναι ότι έχει πλέον προχωρήσει η κατεργασία λιμάτων για την Αγία Πετρούπολη. Σε μεγάλο βαθμό όμως το πρόβλημα που παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα είναι ότι καθυστερεί πολύ η ολοκλήρωσή τους για το Καλίνιγκραντ, παραδείγματι. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. 20 χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία και πάλι με περιορισμένο αριθμό μονάδων και ότι αυτές είναι αρκετά οικονομικές. Και μελετούμε τη στρατηγική για την όλη θαλάσσια ζώνη της Βαλτικής, μια στρατηγική που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2009 με τρεις στόχους, να διαφυλαχθεί η θάλασσα, να συνδεθούν μεταξύ τους οι περιοχές και να εξασφαλιστεί η ευημερία. Υπό την διάσωση της θάλασσας στόχος είναι η καθαρή θάλασσα, τα καθαρά ύδατα στη Βαλτική με τους στόχους για τον περιορισμό των θρεπτικών ουσιών της Συμφωνίας του Ελσίνκη, Η μακροπεριφερειακή στρατηγική ωστόσο δεν προσφέρει νέα κονδύλια. Προσπαθεί να διοχετεύσει τα υφιστάμενα στις μακροπεριφερειακές ανάγκες. Θετικά στοιχεία όπως κύρια προγράμματα που επιτρέπουν και την διάχυση των καλών πρακτικών στην εργασία μεταξύ του περιβαλλοντικού και του γεωργικού τομέα έχουμε εντοπίσει όπως επίσης και σε σχετισμό έχουμε βρει μεταξύ της στρατηγικής και της, ε, του προγράμματος συνοχής στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ε, διαπιστώνουμε όμως ότι η προστιθέμενη αξία της στρατηγικής, προστιθέμενη ως προς τον περιορισμό των, ε, της εισρωής θρεπτικών είναι μια δύσκολη διαδικασία. Διατυπώνουμε προτάσεις, συστάσεις Καταρχάς τα προγράμματα μέτρων θα, υπό την υφιστάμενη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα πρέπει να οδηγούν σε περιορισμό της επιβάρυνσης θρεπτικές ουσίες και θα πρέπει τα μέτρα αυτά να εντοπίζουν τα προγράμματα αυτά να εντοπίσουν πιο αποδοτικά ως προς την ε, οικονομική τους επιβάρυνση μέτρα και μετρήσιμους στόχους περιορισμού των θρεπτικών ουσιών. Τα γεωργικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε ζώνες μεγαλύτερης επικινδυνότητας ορίζοντας ποιες είναι οι πιο ευάλωτες σε σχέση με τα νητρικά ζώνες και στοχεύοντας μέτρα γεωργικά και οικολογικά εκεί που αυτά χρειάζονται περισσότερο και επίσης αποτελεσματικότητα για την ε, διαχείριση των λιμάτων. Θα πρέπει να προχωρεί ταχύτερα στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και να επιτυγχάνει τους στόχους και τη φιλοδοξία της οδηγία, των οδηγίων του 1991 και επίσης θα πρέπει να ε, προγραμματίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η ε, διαχείριση των κλιμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από πλευρά λοιπόν των ελεκτών ε, είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που μα λέτε. Ο κύριο Λερουά λοιπόν τώρα έχει το λόγο. Η κυρία Λερουά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαι σίγουρη ποιο θα πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Μαλγκά, είμαι και είμαι από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που διοργανώσατε την σημερινή συνεδρίαση και εσά και τον εισηγητή αλλά και του προσκεκλημένου μα. Θα σας, μιλά... θα μιλήσω με δύο ιδιότητε. Καταρχάς θα σα παρουσιάσω και την πλευρά τη Helcom, του ε, Σύμβαση για το Ελσίνκι. Μέχρι τον Ιούλιο είμαστε στην ε, Προεδρία τη Helcom και έχω και εγώ προσωπικά την τιμή αυτή. Να ευχαριστήσω καταρχάς λοιπόν ε, το ελεκτικό συνέδριο που παρουσίασε τα ευρήματα του δικαστηρίου, πώς έχουν ήδη εφαρμοστεί κάποιες από τις συστάσεις σας. Ζητώ συγγνώμη, προσπαθώ να βρω τις διαφανίες μου. So, thank you very much. So just this is... Σα σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ βλέπετε λοιπόν ε, ένα σχεδιάγραμμα για το ρόλο των διάφορων ε, ευρωπαϊκών ε, μέσων που συμπεριλαμβάνονται και νομίζω ότι διάφορα από αυτά τα ακούσατε και στην παρουσίαση του Λεπτικού Συνεδρίου να επικεντρωθούμε κυρίως ότι ο ευτροφισμός προκαλείται από το μεγαλύτερη εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από διάχυτες πηγές. Αυτό για την περίοδο 2014 και 2020. Τα κριτήρια ήταν πολύ πιο αυστηρά σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ανάπτυξη τη υπαίθρου. Θα συμφωνήσουμε για την, πολιτική, την κοινή πολιτική αλλά και για την πολιτική συνοχή. Θα είναι ένα εργαλείο που θα δραματίσει μεγάλο ρόλο Κατά δεύτερον, η οδηγία για την εξεργασία των ε, λιμάτων, των αστικών λιμάτων. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ από την ε, δημοσίευση της έκθεσης του Εκτικού Συνεδρίου κάναμε και μια έκθεση υλοποίησης και να σας πω ότι μεγάλη πλειονότητα των κρατών της Βαλτικής συμπεριλαμβανομένων και όλων εκείνων όπου η συμμορφώση ήταν χαμηλή. Ήταν συντόμως σε λίγες εβδομάδες να συμμετάσχετε, συμμετάσχετε σε δημόσιες διαβουλεύσεις ε, για να δούμε κατά πόσον η οδηγία αυτή πραγματικά ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Καλή και χρήσιμη αποδείχτηκε, αλλά θέλουμε να δούμε και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως είπε και ο συγητή στα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν ένα αποτελεσματικό το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Να χρησιμοποιήσω και μία ανεπίσημη, αν θέλετε, έναν επίσημο χαρακτηρισμό. Συνεργαζόμαστε με τον ΩΣΑ, ο οποίος μας βοηθά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσουμε ανάγκε ανάγκες επενδύσεις και τις ικανότητες επενδύσεις θα είναι δυνατή. Άλλα δύο σημαντικά εργαλεία πλαίσιο τώρα. Καταρχάς η οδηγία πλαίσιο για το νερό έχει ολιστική, όπω ξέρετε, συνολική προσέγγιση για όλα τα σώματα υδατός. έχουμε και τις ε, καταστάσεις διαχείρισης. Πίζουμε λοιπόν ότι με τα πορίσματα της αξιολόγησης αυτής θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να διαπιστώσουμε κατά πόσον τα κρατημέλη έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά με την στόχοθεσία, την υλοποίηση κτλ. Και έχουμε και την οδηγία για το αμα, α, και εδώ λοιπόν εξετάζουμε το τι μας αναφέρουν τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση πριν το καλοκαίρι να δημοσιεύσουμε τα πορίσματά μας. Άρα θεωρώ ότι έχουμε ένα σύνολο καινούριων νέων τεκμηρίτης. Ε, ανέφερε σημαντικά κονδύλια. Δεν θέλω να αναφέρω αριθμητικά ποσά, αλλά να έχουμε υπόψη ότι η χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις υγιεινής έχει αντίκτυπο και σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, ούτω καθεξής, όταν μιλάμε για επεξεργασία λιμάτων. Αυτό το τονίζω. Άλλα δύο στοιχεία πρώτη περάσω στην παρουσίαση της σύμβασης του Ελσέκη. Να πω το εξή ότι η οδηγία για τα νετρικά αποδεικνύεται ουσίευσε μια έκθεση για την ε, οδηγία, την εφαρμοστική οδηγία και αυτό λοιπόν θα έχει σημασία και θα πρέπει να το περιμένουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη δεν είναι τα μοναδικά α, κράτη στη Βαλτική. Έχουμε και τη Ρωσία. Η ρωσική επικράτεια αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, πολύ σημαντικότερα από ότι οι γειτονικέ χώρε. Αυτό η Επιτροπή του Ελσίνκη είναι πολύ σημαντικός θεσμικός φορέας. Βλέπετε τις σημαίες των χωρών. Το 1974 παρτιζόταν από ε, χώρες που ήταν τμήματα της Σοβιετικής Ένωσης. Η Γερμανία ήταν ε, διχασμένη τότε. Πάντως ε, η Επιτροπή του Ελσίνκη υπήρχε και στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και βοήθησε και τότε τις χώρες που βρέχονταν από τη Βαλτική να προστατεύουν και πολύ θαρρυντικό που καταλήξαμε σε ομόφωνη άποψη ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να επιταχύνουμε ε, τις δράσεις μας, ε, εφαρμόζοντας τα μέτρα που έχουμε θετήσει και προσδιορίζοντας τις φιλοδοξίες μας για το μέλλον. Και ήταν πολύ σημαντικό και θαρρυντικό, εμψυχωτικό που καταφέραμε και συμφωνήσαμε στο πλαίσιο. Ο ρόλο είναι ένα είδος ε, περιβαλλοντικού συντονιστικού κέντρου, αλλά και φορές χάραξης πολιτικής. Ένα από τα σημαντικότερα πλανεκτήματα της Επιτροπής του Ελσίνκη είναι ότι δημιουργεί ένα φόρουμ για την επιστημονική κοινότητα. Και μάλιστα η Βαλτική είναι πιο προηγμένη περιοχή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Δυστυχώς δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές που έχουν τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία, το ενωσιακό δίκαιο, εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθηκών. Άλλο σημαντικό θέμα από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι καταφέραμε στην Επιτροπή των Ελσιακούς μας στόχους έχει τους ίδιους στόχους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή θέλει να υλοποιήσει καλό μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση για τη Βαλτική την επόμενη δεκαετία. Σε ό,τι αφορά τον ευτροφισμό, όπως ε, θα ακούσετε και αργότερα και φαντάζομαι οι εμπειρογνώμενες είναι σε καλύτερη για τη Βαλτική και ε, βλέπουμε ποια είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες εισρωές τρεπτικών ουσιών ε, φυσικά συμβαδίζοντας με τα επιστημονικά πορίσματα για το τι είναι εφικτό. Δεν σας αναφέρω λεπτομερώς τα στοιχεία αυτά, πάντως μπορούμε να περάσουμε στους δεύτερους στόχους που είναι ε, μια προσέγγιση ελέγχου των εκπομπών. Εν κατακλείδη πάντως ε, ε ακόμη μαθαίνουμε από τις προτάσεις αυτές και είναι πολύ ενδιαφέρον πείραμα για το ποια θα είναι η ακολουθητή απορία για τα κράτη-μέλη και στο μέλλον. Και κάποια σχετικά θετικά νέα. χρησιμοποίησαμε κάτι, κάποια πιο επικαιροποιημένα στοιχεία με τις δύο τελευταίες χρονιές και διαπιστώνουμε μείωση 24% του φωσφόρου και 22% μείωση του αζότου. Κάτι πολύ θετικό στην περίοδο 1995 μέχρι το 2014 και για να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στην ίδια περίοδο το ΑΕΠ των περισσότερων, για να μην πω όλων των χωρών γύρω από τη Βαλτική, σημείωνε μείωση. Είναι σημαντικό λοιπόν που ε, κατέστη δυνατή μείωση των, του φωσφόρου και του αζότου παρόλο που η αύξη, υπήρξε αύξηση της οικονομικής ε, δραστηριότητας. Στη συνέχεια οι εμπειρογνώμονες θα εγκύψουν σε πιο επιστημονικά θέματα και πιο επιστημονικές σκοπιές, αλλά από την άποψη της χάραξη πολιτικής διαπιστώνουμε ότι θεσπίστηκαν κάποια μέτρα, αλλά ίσως δεν είναι αρκετά ευρεία ε, και ίσως ε, χρειάζεται χρόνος για να αποφέρουν αποτελέσματα. Και δεν το χρησιμοποιούμε αυτό μόνο δικαιολογία ως πρόσχημα. Και φυσικά υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που ανακύπτουν και που συμβάλλουν στον ευθροφισμό. Ενίσχεται η οξύνηση λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού στη θάλασσα και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Επίσης, το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε ομόφωνα από τους εταίρους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Έχουμε βέβαια ακόμη λίγα χρόνια στη διάθεσή μας, οπότε Προσπαθώ να είμαι κάπως αισιόδοξο, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο. Και εδώ έχετε ένα πίνακα. Στο άνω τμήμα βλέπετε τις κοινέ δράσεις, τις, δράσεις, τις δράσεις δηλαδή που συμφώνησαν να διεκπαιρεώσουν από καινού οι χώρες. Τα γαλάζια είναι τα καλά νέα, τα κίτρινο τμήμα είναι το πιθα... δυνητικά καλά νέα και το κόκκινο τμήμα είναι... δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα, δεν έχει εφαρμοστεί η δράση και άρα ακόμη δεν έχουμε καλά νέα. Πιο κάτω βλέπουμε κάπως πιο αρνητική εικόνα, τις εθνικές δράσεις, τις δράσεις λοιπόν που ίδιες οι χώρες ε, πρότειναν να αναλάβουν για να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του ευτροφισμού. Βέβαια, θέλουμε να έχουμε μια γενική επισκόπηση ε, ότι ο ευτροφισμός περιλαμβάνεται στους κοινούς στόχους. Βέβαια, οι κοινέ δράσεις ε, έχουν υλοποιηθεί, αλλά οι εθνικές δράσεις για την καταπολέμηση του ευτροφισμού δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί στους Γιατί κάποια απλά και σχετικά ε, φθηνά, ε, φθηνά πράγματα έχουν γίνει. Δεν χρειάζεται να είναι δαπανηρά για να έχουμε αποτελέσματα. Βέβαια κάποια μέτρα γίνονται όλο και πιο δαπανηρά. Για παράδειγμα, κάποια μέτρα που έγιναν εφαρμόστηκαν από τα λύματα. Επίσης, δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνικό και επιστημονικό. Είμαστε σε επίπεδο χάραξη πολιτικής, πολιτικό. Πάντως αναλύουμε την αποτελεσματικότητα και των εθνικών μέτρων. Πάντως είναι σημαντικό ε, να κάνουμε μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων για να δούμε ποια θα είναι η ακολουθητέα ανάλυση που έκανε η Επιτροπή του Ελσίνκη. Και βλέπετε τις ε, εκτιμήσεις για τις αιτήσει ε, ζημίες από τον ευτροφισμό που είναι της τάξης των 4 δισεκατοντική και άποψη ψυχαγωγική, από απώλεια ευκαιριών δηλαδή και από την αποτελμάτωση κατάσταση, από την έλλειψη βελτίωσης. Αυτά σας ευτυχεί όσο περισσότερο γίνεται, ενώψη και της πιθανότητα οι κλιματικές αλλαγές να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά. Σήμερα κοιτάμε πάλι προς τα μπρος, κοιτάμε να δούμε τι έχουμε επιτύχει, γιατί αυτά που δεν επιτύχαμε δεν τα επιτύχαμε. Για το προσεχές πολιτές νομικό πλαίσιο, τους προσεχείς κανονισμούς. Γι' αυτό και θέλω να μου απαντήσει 12 μέχρι το 14 γιατί, γιατί η κατάσταση είναι τέτοια Δεν θα ήταν δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα ε, ε, πιθανό και πολύ δύσκολο να το εξηγήσει κανείς αυτό στον πολίτη και ψηφοφόρο ανεξαρτήτως οι άλλες είναι το 2000 και το 2008. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τη δυσφορία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Πρόεδρος, ναι, θα κάνω και εγώ κάποια ερωτήσει, ευχαριστώντας για τις πολύ ενδιαφέρουσε εισηγήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα και ποια είναι αυτά. Και δεύτερον, σε σχέση με την ε, Ρωσία και την συμμετοχή στη σύμβαση. Ρωσία και Λευκορωσία. Γιατί βέβαια είναι απαράδεκτο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθούν να περιορίσουν ε, το φαινόμενο και να, έχουν, ε, να τηρούν τους όρους της Λευκορωσία. Γιατί βέβαια είναι απαράδεκτο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθούν να περιορίσουν ε, το φαινόμενο και να, έχουν, να τηρούν τους όρους της σύμβασης, ενώ η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν το πράττουν. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν εδώ και δεύτερο, κύριος Σαουάρμα, ειδικά για την Πολωνία. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο τα μέτρα, και ήταν πολλά, το είδαμε, υπήρξαν και ε, κατασκευές μονάδων καθαρισμού λιμάτων κτλ. Γιατί δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα. Μάλιστα ρωτώ από τις στιγμή θα σταματήσουν να μπαίνουν νέες τρεπτικές ουσίες, επιβαρυντικές τρεπτικές ουσίες. Προς την Επιτροπή βεβαίως. Απάντηση, ναι, ευχαριστώ πολύ. Όντω είναι δύσκολε ερωτήσει. Αλλά γι' αυτό με πληρώνετε. Για να δίνω καλέ απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ με την τελευταία σας ερώτηση που θα δυσκολευτώ πιο πολύ. Ελπίζω οι, οι άλλοι δύο συναδελφοί να έχουν καλύτερες απαντήσεις. Πάντως, με απόλυτες συνέπειες της ε, υπερπαρουσίας τρεπτικών ουσιών έχουμε από την Υπουργική Συνεδρίαση διαπίστωση ότι κατά 95% η Βαλτική είναι επιβαρημένη ως προς τις λεγόμενες θρεπτικές ουσίες. Είναι ρηχή θάλασσα, έχει δηλαδή φυσικές συνθήκες. Οικονομικά έχει δραστηριότητα αιώνων, έντονη δραστηριότητα αιώνων, μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και είναι ένα γεγονός αυτό της επιβάρυνσης το οποίο δεν μπορούμε να αποκρύψουμε. Άρα είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε είναι κάποια ακολουθήση, τουλάχιστον σε σχέση με την οδηγία για, το θαλάσσιο περιβάλλον. Βλέπουμε το σύνολο, δηλαδή ξέρουμε ότι ο ευτροφισμός επηρεάζει και τη γονιμότητα των ε, ηχθείων, ε, ότι δεν θα είναι τόσο παραγωγική όλη η περιοχή κτλ. Ταυτόχρονα όμως κοιτάμε να δούμε σε όλα τα μέτωπα τι μπορούμε να κάνουμε, να μειώσουμε και ούτω καθεξής και προσπαθούμε να δώσουμε μια πιο. και αυτή είναι η γενική απάντηση που μπορώ να δώσω. Μπορώ να δώσω μια πιο ολιστική προσέγγιση. Και βέβαια στην ερώτηση τι κάνουμε καλύτερα, αν κοιτάξουμε προ τα πίσω κτλ. Κοιτάξτε, πάντα εξαρτώμεθα από το τι έχουμε πίσω μα. Κοιτάμε εκθέσει, τουλάχιστον δύο-τρει εκθέσει δεδομένα. Αλλά και όπω είχα απαντήσει άλλωστε και το 2016, αυτό που κάνουμε είναι ότι όλοι οι φορείς υιοθετούν από κοινού προγράμματα, κανόνες, οι κανόνες παραδείγματι για τη χρηματοδότηση, πρόγραμμα ε, ανάπτυξη πέθρου που αναφέρατε κι εσείς, έχουν συγκεκριμένους στόχους ε, μεταξύ των Έχω συνείδηση του γεγονότος ότι και όντως έχουμε λάβει υπόψη και το λαμβάνουμε πάντα υπόψη, ε, το τονίζουμε προς πάντα ενδιαφερόμενο τι είδους διαπιστώσεις έχουμε στα χέρια μας πάντα ενημερώνουμε. Είναι συζήτηση με τα λόγου γνώσεως και δεν ξέρω αν θα ακουστεί πολύ διπλωματικό αυτό που λέω, ε, έχουμε εδώ τις συνέπειες της οικονομικής δραστηριότητας και της παρουσίας της ανθρώπινης πληθυσμιακής ε, ε, πυκνότητας που έχει η περιοχή. Μας να κάνουμε το μερίδιο της δουλειάς μας αναλογή, να αναπτύσσουμε θετικές δραστηριότητες, να ορίζουμε προϋποθέσεις για κάποιες δραστηριότητες που θα είχαν αρνητικές συνέπειες και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο φιλόδοξη πρόοδο από ό,τι αν ο καθένα έμενε στη γωνιά του. Και αυτό το λέω για να κάνουμε τη σύγκριση με την κατάσταση πριν από 15 χρόνια, η οδηγία παραδείγματι για τα αστικά λύματα. 12 ε, κράτη-μέλη, 12 νέα κράτη-μέλη ε, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόοδο πολύ ταχύτερη σε αναλογία κλίμακας έναντι αυτής που είχαν τα προηγούμενα κράτη-μέλη στην προηγούμενη 15 ετία. Είχαν όμως τεράστιες ανάγκες σε επενδύσεις για εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηριστικά τοπική λειτουργία. Όσα όχι μόνο για την εκπλήρωση των στόχων των περιβαλλοντικών, αλλά ταυτόχρονα και των ρυθμών, για να βελτιώσουμε τους ρυθμούς της υλοποίησης. Τίποτα άλλο από μια ειλικρινή απόπειρα να δώσω απαντήσει, δεν μπορώ να προσφέρω δευτερόλεπτα για να συζητήσω με τη συνάδελφο. Ίσως είναι προτιμότερο να το ξανακοιτάξουμε και να περιμένουμε να ξανάρθει η σειρά μας ή να σας στείλουμε και ένα mail, γιατί είναι απαραίτητο να σας δώσουμε ακριβείς πληροφορίες, κυρία Νίμεν, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Η μείωση των θρεπτικών ουσίων δεν θα εκδηλωθεί αυτό καλύτερα, σε καλύτερο περιβάλλον απαραίτητα. Εδώ ο συνάδελφο μπορεί να μα εξηγήσει κάπω καλύτερα τι εργασίε λοιμάτων. Πραγματικά ε, συνάδουν με τι ε, και τα πρότυπα τη Σύμβαση του Ελσίνκη και τη Επιτροπή του Ελσίνκη. Και η επιστημονική κοινότητα το επιβεβαιώνει αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τι και εμπόδιο στην στοχοθεσία, στη στοχοθέτηση των μέτρων. Άρα υπάρχουν υπάρχουν και κατά. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, πραγματικά, ένα σημείο το οποίο επιδέχεται βελτίωσης. Ευχαριστώ. Να παρουσίασαν ένα master plan, όπως ονομάστηκε, ένα κεντρικό σχέδιο, ένα σχέδιο λεπτομερές για τις επενδύσεις και για την υλοποίηση. Έχει γίνει μία σημαντική μεταρρύθμιση της διαχείρισης. Έχουν, θα πετύχουν δηλαδή καλύτερα αποτελέσματα και θα επιταχύνουν την ανταπόκριση. Για την ερώτηση που κάνατε για τα βασικά και η Ρουσία έχει πετύχει τους στόχους ότι αφορά Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ή θα πρέπει να εξεταστεί ως υπολεκάνη. Και σε κάποιες περιπτώσεις... Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία συγκεκριμένα ανά ε, και αναπεριοχή, θα θέλαμε να τα έχουμε αν μπορείτε να μας τα χορηγήσετε. Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της ε, παρουσίασης από την, ε, το Πανεπιστήμιο της Ομπορκ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, μου ζητήσετε να κάνω μια επισκόπηση των ε, αναγκών σε ό,τι φορά την καταπολέμηση του ευστροφισμού στην περιοχή της Βαλτικής. Καταρχήν να σας πω από πού έρχομαι και τι ρόλο έπαιξαν οι επιστήμονες στην παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή του Ελσίνκη και τι είδους έρευνα κάναμε στη Βαλτική σε ό,τι αφορά τον ευτροφισμό. Στη συνέχεια θα σας πω δύο λόγια για μερικά θεμελιώδη ζητήματα, δηλαδή και όπως η χρηματοδότηση, θα δούμε πώς λειτουργεί και εμείς έχουμε λάβει σχετική χρηματοδότηση για έρευνα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ευτροφισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κονδύλια και θα σας δώσω κάποια αποτελέσματα εν συντομία. Θα δούμε τι γνώσεις ε, συγκέντρωσε η παρήγαγη επιστήμη της αιτής ε, του ευτροφισμού στις λεκάνες απορροής, ε, ποια είναι τα αποτελέσματα στα υδατικά συστήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις ε, ε, στα νυχτά της Βαλτικής και θα σας δώσω και κάποιες συστάσεις. Καταρχήν, προέρχομαι από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, από το Κέντρο για τη Βαλτική Θάλασσα. Έχουμε, κάνουμε έρευνα για το θέμα αυτό. θα σας ενημερώσω γι' αυτό αργότερα και μάλιστα έχουμε και το Ινστιτούτο της Βαλτικής, Baltic Nest και εμείς κάναμε τους υπολογισμούς, τους επιστημονικούς υπολογισμούς για το τι θρεπτικές ουσίες θα πρέπει να αφαιρεθούν, να απομακρυνθούν από ποια χώρα, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ότι οι επιστήμονες συνεργάστηκαν πολύ στενά μαζί με την Επιτροπή του Ελσίνκη και με τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Και είναι πολύ θετικό που επιτέλους υιοθετήθηκαν τα επιστημονικά πορίσματα και έγιναν δεκτές οι επιστημονικές ε, συμβουλές. Και αυτό ίσως θα είναι καθοδήγηση για τις μελλοντικές στρατηγικές για τη Βαλτική ε, σε σχέση με άλλε λεκάνες όπως της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και ούτω καθεξής. Ε, θα σας μιλήσω και για το θέμα το, της επικοινωνίας. Έχουμε εδώ μια ομάδα, το Baltic Eye, σε συνεργασία με δημοσιογράφους, με πολιτικούς ηθήνοντες και ασχολούμαστε με, την, με την, τον ευτροφισμό, την βιοπικιλότητα και το πώς επηρεάζεται η αλία στη Βαλτική. Έχουμε επίσης κάποια φυλάδια πολιτικής που ασχολούνται με το θέμα του ευτροφισμού στη Βαλτική και μάλιστα τα έχω φέρει μαζί μου. Μπορώ να σας τα δώσω ή να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για την καταπολέμηση του ευτροφισμού. Ε, έχουμε μια σύνοψη των μέτρων ε, που περιλαμβάνονται σε αυτά τα εγχειρίδια της πολιτικής. Αυτά ως προς το υπόβαθρο για να δείτε από πού προέρχομαι και τι ρόλο παίζει το Ινστιτούτο μας ε, στα θέματα του ευτροφισμού στη Βαλτική. Όπως είπα και προηγουμένως, ο ευτροφισμός προκαλείται κυρίως από την εισρωή ε, θρεπτικών ουσιών από τη γη προς την θάλασσα, από άζωτο, φόσφορο κυρίως, κάτι που προκαλεί έξαρση φυτοπλακτού. Και πριν η πρόεδρος ρώτησε, γιατί ε, το σύστημα αντιδρά τόσο αργά. Γιατί έχουμε ένα στενοπό στο κάτεγκα της Κάγκερακ και με αποτέλεσμα ε, να έχουμε πολύ αργή ε, και παραμονή μάλλον στις λεκάνες αυτές. Οπότε δεν έχουμε διάλυση όπως άλλους, σε άλλες υδάτινες λεκάνες. Χρειάζονται 30 χρόνια για να διαλυθούν αυτές οι θρεπτικές ουσίες. Επίσης, ε, είναι χαμηλή η ισορροή προ το, ε, του φρέσκου ύδατο και δεν έχουμε αρκετό οξυγόνο στην Βαλτική που έχουμε, και έχουμε μεγάλες περιοχές χωρίς οξυγόνο, ανοξυγονικές. Ε, σε περιοχές χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχει δυνατότητα ζωής. δεν έχουμε μύδια, δεν έχουμε ανώτερη ζωή. Ε, δεν έχουμε οστρακοειδή, δεν υπάρχουν ε, ε, αλλιεύματα σε αυτές τις ανοξυγονικές ζώνες. Και μάλιστα εξαπλάστηκαν έως δεκαπλασιάστηκαν αυτές οι ανοξυγονικές ζώνες τα τελευταία χρόνια. όλα αυτά τα συζητούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο δράση για τη Βαλτική που είναι πολύ φιλόδοξο σχέδιο δράσης και μάλιστα εδώ έχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, θέλουμε καθαρότερο νερό στη Βαλτική, γιατί καθαρότερο νερό σημαίνει λιγότερα φύκια, λιγότερο φυτοπλακτό, λιγότερες θρεπτικές συνθήκες και καλύτερες συνθήκες βιοπικιλότητας. Συμφώνησαν οι εμπειρογνώμονες ε, στο Helcom για τα θέματα αυτά και με κάποια αμερικανικά μοντέλα προσπαθήσαμε να αποσυντικοποιήσουμε τους στόχους, δηλαδή τι αφαίρεση θρεπτικών ουσιών πρέπει να πραγματοποιήσει κάθε χώρα, τι απομάκρυνση πρέπει να πραγματοποιήσει κάθε χώρα. Αυτή είναι η συμβολή της Helcom σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, είναι πολύ ευάλωτο το θαλάσσιο σύστημα της Βαλτικής, πολύ πιο ευάλωτο από άλλα υδάτινα συστήματα και αυτό είναι το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά ε, τη χρηματοδότηση, είχαμε το σχέδιο Bonus που εγκαινιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 185 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά τα ακρονίμια. Πάντω, 50% των κονδύλιων προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από εθνικά κονδύλια. Γενικώ είχαμε 100 εκατομμύρια ευρώ συνολικές δαπάνες για έρευνα στη Βαλτική θάλασσα. Και μάλιστα στη γραμματεία του Μπόνου στο Ελσίνκι ε, ζήτησα κάποια στοιχεία και πήρα τα εξή. Γενικώ 34 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε έρευνα στη Βαλτική θάλασσα για τον ευτροφισμό. Ένα τρίτο του συνολικού ποσού μπορεί να θεωρείται μεγάλο το ποσό, αλλά μιλούμε για 10 χρόνια, για 8 χρόνια συν τη Ρωσία. Γιατί και η Ρωσία μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Bonus. Και μάλιστα είχαμε πολύ καλή συνεργασία με Ρώσου εμπειρογνώμονε. Μερικέ φορέ είχαμε προβλήματα για τη συμμετοχή του γιατί δεν χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προσετεριστούμε και του ε, Ρώσους εμπειρογνώμονε. γιατί η Ρωσία είναι σημαντικός ε, στη Βαλτική και ήταν σημαντικό να συμμετέχει. Ω προ τα αποτελέσματα, έχουμε ξαναδεί αυτά τα στοιχεία. Βλέπετε εδώ την εικόνα του, της λεκάνης απορροής. Και αυτή είναι η αιτία του ευτροφισμού. Η κίτρινη περιοχή είναι οι καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις. Ε, Γερμανία, Πολωνία, Δανία, χώρες της Βαλτικής, στη βόρεια στο βόρειο τμήμα έχουμε λιγότερο, Γεωργία, λιγότερο από 10%. Πολωνία, Γεωργία, ε, Γερμανία έχουν 60% της επιφάνειας ε, ε, γεωργικές εκτάσεις. Οπότε κυρίως η Γεωργία ε, συγκεντρώνεται στη νότια περιοχή. Και έχουμε κάποιες πιο μακροπρόθεσμες ε, μακροπρόθεσμους υπολογισμούς στις ουσίες από τη δεκαετία του 80 και έγινε κάποια μείωση, αλλά το θέμα είναι ε, ποιο είναι το, ο ελέφαντος στο δωμάτιο, γιατί είναι τόσο αργή η διαδικασία. Το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό. Βλέπετε ε, ένα πίνακα με τις εισρωές ε, των θρεπτικών ουσιών στις λεκάνες απορροής. 7 εκατομμύρια τόνοι αζότου και φωσφόρου μπαίνουν στις λεκάνες απορροής. Βλέπετε τα εξωτερικά βέλη και όσο μπαίνουν στη λεκάνη απορροής, μαζί με τα λοιπάσματα, τις ζωοτροφές, τις τροφές, μπαίνουν λοιπόν στη λεκάνη απορροής και 70% όλων των καλλιεργιών που καλλιεργούνται στην, στη λεκάνη απορροής της Βαλτικής, από όλες τις χώρες δηλαδή που, που παράγουν κρέας, που έχουν κτηνοτροφία. Αυτό είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Ε, αυτό, αυτό δημιουργεί το πρόβλημα του ευτροφισμού. Οι μεγάλες εισρωές λόγω της κτηνοτροφίας. Και αν δεν το περιορίσουμε, θα επιδεινώνεται η κατάσταση στη Βαλτική, που έχει πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Και μάλιστα η κτηνοτροφία στη Βαλτική έχει τριπλάσια παραγωγή ε, κοπριάς και παραγωγή άρα αζότου και φωσφόρου από ό,τι τα αστικά λίματα. Η κτηνοτροφία λοιπόν είναι ο ένοχος, ο βασικός. Και έχουμε μια πολιτική που, παραγωγής ε, κοπριάς που δεν ξέρουμε πώς να την απομακρύνουμε, πώς να, που να την διοχετεύσουμε. Βέβαια έχουμε τεχνικές για τη μεταφορά της κοπριάς, τη ε, της εφαρμογής των λιπασμάτων, δεκαπλασιασμό της χρήσης λιπασμάτων από τη δεκαετία του 60. Το γαλάζιο τμήμα είναι αν μόνο το φωσφόρο σαν μια πόλη 300.000 χωρίς αποχέτευση. Η κτηνοτροφία λοιπόν είναι ο υπέτειος ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Επίσης, αναφέρθηκε προηγουμένως η Δανία. Εκεί η αποθήκευση της κοπριάς είναι μια τεχνική που μπορεί να αποφύγει κοπριά, να τη μετατρέψουμε σε λίπασμα, να δημιουργήσουμε ζώνες ανάσχεσης. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε το διαρθρωτικό πρόβλημα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει επιτύχει η Δανία. Ε, έχουμε 6 εκατομμύρια δανούς με παραγωγικές εστίες και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ποιες είναι οι περιοχές στόχοι και αυτό είναι γνωστό για τη Δανία αλλά όχι για όλες τις ε, άλλες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα. Και ε, ερχόμαστε στα παράκτια ύδατα. Εκεί έχουμε κάποια θρεπτικών ουσιών από τους σταθμούς επεξεργασίας ε, στα αστικών λιμάτων. Αλλά βλέπουμε εδώ για τα μύδια ε, και άλλα ε, θαλασσινά που λειτουργούν ως φίλτρα και καθαρίζουν το νερό, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα συστήματα. Πάντως, είδατε αυτά τα, το φυτοπλακτόν τα κυανοβακτήρια και αυτή η έξαρση φυτοπλακτού που διαπιστώνουμε κάθε καλοκαίρι. Βέβαια και αυτά τα, τα φύκια έχουν ένα ρόλο στο, στον κύκλο, γιατί όσο αυξάνεται βέβαια η θερμοκρασία, αυτό είναι τροφή για τα αλλιεύματα και ίσως έτσι αυξηθούν ε, τα αποθέματα ρέγκασης ή με την αύξηση των φυκιών. Τώρα τα θέματα παρακαταθήκης ε, σε ό,τι αφορά τις θρεπτικές ουσίες. 30 χρόνια στη Βαλτική χρειάζονται για Και έχουμε περάσει βέβαια από φάση υπερβολικής συγκέντρωσης των θρεπτικών ουσιών σε φάση ε, απεμπλουτισμού. Και στην κυρίως Βαλτική έχουμε αργή μείωση της συγκέντρωση. αλλά θα χρειαστούν 20 με 30 χρόνια για την καθάριση. Αυτό είναι πω στη λεκάνη απορροής είναι το πρόβλημα. Στη Σιλεσία, στη, στη, στην Πολωνία ή στις ακτές της Πολωνίας, για να ξέρουμε πού θα επικεντρώσουμε την έρευνά μας. Επίσης, δεν έχουμε μέχρι στιγμής δυναμικά μοντέλα για να δούμε τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μέτρων. Γνωρίζουμε ότι η κοπριά είναι ο βασικός ένοχος, αλλά θα πρέπει να βελτίωση της κατάστασης στη Βαλτική. Για τα παράκτια ύδατα, η βιοπικιλότητα και η λειτουργία των οικοστημάτων δεν περιγράφονται επαρκώς. Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων, να δούμε τη στάθμιση μεταξύ της γαλάζιας ανάπτυξης και των ε, υπηρεσιών οικοσυστημάτων και σε πλακτού στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε όμως και την παρακαταθήκη του, ε, των θρεπτικών ουσιών άνθρακα στα ειζήματα η χρηματοδότηση του προγράμματος Bonus, που ήταν πολύ σημαντική για την έρευνα και μάλιστα ήταν πολύ επιτυχημένο σχέδιο, φτάνει στο τέρμα τη. Βέβαια, υπάρχει μια πιστεύω και νομίζω ότι εδώ εκπροσωπώ όλη την επιστημονική κοινότητα ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη μια τέτοια παράταση και αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης ε, ε, και συνδυασμού ευρωπαϊκών κονδυλίων και εθνικών κονδυλίων ε, έχει θετικά αποτελέσματα. Και τέλος, την που είμαι πολιτικός, κανένας επιστήμονας ποτέ δεν με πλησίασε για να μου παρουσιάσει τα πορίσματά του. Γι' αυτό και θα πρέπει να εκλεκεύσουμε περισσότερα τα πορίσματα της επιστήμης και να τα φέρουμε πιο κοντά στην πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ε, τουλάχιστον εμείς τα καταλάβαμε εδώ πέρα και αν δεν αλλάξει τίποτα. Για ότι μετατρέπεται σε, σε στερεά, σε γη. Όχι, ευτροφισμός δεν σημαίνει ότι θα ξεραθεί όπως μια λίμνη, ότι θα υπάρχει δηλαδή κόρπινα. Φιλανδικό Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Στην παρουσίαση αυτή θέλω καταρχάς να δώσω μια επισκόπηση του ευτροφισμού και να αναφερθώ και στις διάφορες τάσεις εισρώων και μέτρα που έχουν μέχρι τώρα εισαχθεί με αξιολόγηση της επιτυχίας τους ή όποιων στοιχείων έχουν σχέση με την επιτυχία τους. Λέγεται μερικές φορές ότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι επιστήμονες. Εγώ όμως ε, συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Ήταν πολύ καλές οι παρουσιάσεις. ε, πάσει από ευτροφισμό η Βαλτική θάλασσα, σωστό αυτό. Πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση, πρόκειται για κάτι το καινοφανές. Έχουμε συνάντηση της Helcom στην Λιθουανία για να δούμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ευτροφισμού. Εδώ βλέπετε μόνο τα χωρίδατα της Φινλανδίας στο χάρτη ε, μερική εικόνα, αλλά το ίδιο ισχύει σε όλη τη Βαλτική. Το κόκκινο σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα περιβαλλοντικά. Ωστόσο, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε ακολουθεί διαφορετικούς δείκτες, διαφορετικά είδη δικτών και έτσι αν είχαμε άλλους δείκτες θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε τη βασική πανίδα με το πράσινο σε καλή κατάσταση, βασική πανίδα, βενθική πανίδα ουσιαστικά και όπου βλέπετε πράσινο, πράσινο σημαίνει καλές ε, συνθήκες. Και μετά βλέπετε το φυτοπλανκτόν και τη χλωροφύλη, δείκτες που δείχνουν κακό επίπεδο σε όλες τις, ε, σε κάθε σημείο των εγχώριων υδατών της Φιλανδίας, σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Επομένως, οι λοιποί δείκτη βρίσκονται κάπου μεταξύ των χρωμάτων που βλέπετε. Λέγεται ότι μια τέτοια κατάσταση αργεί να ανατραπεί. Έχουν γίνει και αναφορές στις σχετικές έρευνες. Ε, ωστόσο κάποιες βελτιώσεις βλέπουμε και κυρίως έχουμε να κάνουμε με τη ρίζα ε, της εισρωής των θρεπτικών ουσιών. Αυτό κοιτάμε εδώ και εδώ βλέπετε στα αριστερά περιορισμό των αζώτων, αζωτούχων ενώσεων και δεξιά των φωσφόρων σε διάφορες υπολεκάνες της Βαλτικής. Όσο πιο μεγάλο είναι το σήμα που βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη και η μείωση των ε, αιτίων ε, εισρώων. Στον φόσφορο συγκεκριμένα, δεξιά βλέπετε τον κόλπο της Φιλανδίας, τον φιλανδικό κόλπο, με μείωση 50% για την περίοδο 97-2003 και 12-14. Βλέπετε επίσης σημαντική μείωση σε κάθε υπολεκάνη πλην του κόλπου της Ρήγας που τη βλέπετε σε χρώμα καφέ κάτω δεξιά. Στη συνέχεια βλέπετε πιο ε, μεγάλους χρονικούς ορίζοντες και την εισρωή θρεπτικών ουσιών στη δεκαετία του 60, του 70, του 80, ακόμα και του 90 είχαμε ριζική αύξηση. Και μετά ήρθανε οι συστάσεις της Helcom και τα ε, νέα μέτρα που οδήγησαν σε σημαντική μείωση, αν και ακόμα δεν έχουμε φτάσει, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, ε, στους στόχους μας. Εδώ έχετε ένα καλό παράδειγμα που εξηγεί και το γιατί ήταν τόσο μεγάλη η μείωση των φωσφορούχων ενώσεων στον κόλπο της Φιλανδίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την μονάδα ε, καταργασίας λιμάτων της Αγίας Πετρούπολης που ξεκίνησε να λειτουργεί από τις αρχές δεκαετίας του 2000 μέχρι πρόσφατα έχουμε τη μέτρηση με πολύ καλή επιτυχία που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απολύτως, τη μείωση στην ε, παρουσία φωσφορικών ενώσεων στον φιλανδικό κόλπο. Εδώ βλέπετε εγκαταστάσεις που αποτελούν πηγές, σημειακές πηγές ε, αποβλήτων φωσφορικών που εισραίουν στην θάλασσα με τη μονάδα κατεργασίας που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καθαρισμό και έτσι διαπιστώθηκε, έγινε μία μέτρηση των αποθεμάτων σε φόσφορο που είχαν καταληφθεί σε προηγούμενες περιόδους και έγινε η μέτρηση της διαρροής φωσφόρου από αυτό. Και έτσι είχαμε μια σημαντική μείωση σε σχέση με, την, ε, εισερχόμενη, με τις εισερχόμενες ποσότητες. Σε τίσους όρους έχουμε 20% μείωση σε βιολογικά διαθέσιμο φόσφορο. Με μία μόνο μονάδα. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν ε, το να μπορούμε στις ε, ε, σημειακές πηγές να βελτιώνουμε την κατάσταση. Και βεβαίως Υπάρχουν δύο δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε με δύο αποθέματα αποβλήτων σε φωσφορικό γύψο στην Πολωνία που οδηγούν σε μεγάλη συγκέντρωση στις παραποτάμιες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αυτά και βεβαίως έχουμε και ε, αστικά κέντρα με σημαντική παρουσία αζότου που θα μπορούσε ευχερός να απομακρυνθεί. Και αυτό βεβαίως αφορά και περιοχές δυτικής, ε, βόρειο-δυτικής Ρωσίας όπου είναι λίγες οι μονάδες καθαρισμού λιμάτων με περιορισμένα αποτελέσματα. Η εισρωή από, τους, ε, από των ποταμών βεβαίως είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία από τον ποταμό Ντάουγκαβα που εισραίει στη Βαλτική, στο ύψος της Ρήγας και άρα θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Όταν μιλούμε για οι ελώδεις περιοχές, οι οι ζώνες ανάσχεσης ε, έχουν περιορισμένο μόνο ε, εκτεταμένοι. Άρα οι μόνοι περιορισμοί που διαπιστώνουμε ήταν αυτοί που αποδίδονται στον περιορισμό, την, ε, για τον περιορισμό των, για την αφαίρεση των από τη θάλασσα με εκτιμήσεις κόστους ανακυλό φωσφόρου. Ε, μια υπόθεση που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε θα ήταν αυτή των ε, ε, υλικών με βάση το ασβέστιο που της περιεκτικότητας σε φόσφορο χάρη στην μέθοδο αυτή με κόστος κατά ένα τρίμα στα δεξιά ηχθείο καλλιέργειες σε κλωβούς μέσα στο νερό συνήθως, στη Βαλτική, καμιά φορά ακόμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το ερώτημα όμως είναι μπορούμε μια στρατηγική τέτοιου τύπου να τη στηρίζουμε σε μια πεπαλαιωμένη ε, και για να ολοκληρώσουμε τα συμπεράσματά μου, τα οποία είναι πολύ απλά. Πρώτον, καλύτερα, καλύτερη απόδοση στους Έχουμε το μεγαλύτερο βάρος, το μεγαλύτερο φόρτο που θα είναι και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αλλά υπάρχουν κάποιες μέθοδοι και πρέπει επίσης να μιλισμονούμε ότι κατά τα χρόνια αυτά της περιβολικής χρήσης των λοιπασμάτων έχει χρειάστηκε να απαντήσει ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Αναλαμβάνω εγώ τα καθήκοντα του Προεδρεύοντος, δίνω το λόγο στον εαυτό μου, για όλες τις πρακτικές πτυχές του νομοθετικού έργου. Και ο κ. Χουμπολκ και ο κ. Κόρμπιν να μας πούν το εξή. ποια θα ήταν τα τρία κορυφαία στοιχεία τα οποία θα βάζατε στην νομοθετική διαδικασία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ελέγξουμε. Κοιτάξτε, δύο θέματα υπάρχουν. Το θέμα της κοπριάς δεν είμαι ειδικό, ε, αλλά σε θέματα τέτοια αντιμετωπίζω. Θεωρώ ότι χρειάζεται πιο μεγάλη ισορροπία να υπάρχουν και οι δύο πτυχέ ε, και η κοπριά και τα άλλα μεταθέσιμε. Μπορεί να γίνει μεταφορά τη κοπριά. Γίνεται στην Ολλανδία, στη Γερμανία, 40-50 χιλιόμετρα παραπάνω. Δεν έχει νόημα από πλευρά. Ε. Υπάρχουν και διαφορετικέ όμω λύσει οι οποίες θα πρέπει να προτιμηθούν. Και κατά τρίτον, θεωρώ ότι ακόμα μπορούν να γίνουμε πολλά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κορμίνα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Είναι δύσκολο να προσθέσω και άλλα τρία μέτρα, πέρα από αυτά που ανέφερε ο συναδελφό. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε προηγουμένω για τι ε, σημειακέ πηγές. Όλες οι χώρες στην Βαλτική μπορούν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την κατάσταση. Και στο Βορρά, στα Φιλανδία και στη Σουηδία μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, επεξεργασία ε, των εσωτερικών υδάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα... το άζωτο. Η γεωργία, ΑΜΒ, η οποία η βασική πηγή των θρεπτικών αυτών ουσιών δεν ε, εκπροσωπείται, δεν αντιπροσωπεύεται όσο θα έπρεπε. Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μια βελτίωση σε ό,τι αφορά το χώρο της Βαλτικής. Και θα ήθελα να προσθέσω, αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα ανακύκλωση στο σύστημα της Γεωργίας, θα μπορούσαμε σχεδόν, σχεδόν ε, να υλοποιήσουμε το να διαπιστώσουν, θα πρέπει να διαπιστώσουν και ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τους ε, κατηγορήσουμε. Θέλουν υποστήριξη από την τροπημένη καλλιέργεια. Η πρόεδρο τροπημένη καλλιέργεια. Η πρόεδρο τι αφορά την ε, διάχυση θρεπτικών ουσίων στις ε, αγωγούς. Τι λείπει το νερό αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα στη γεωργία. Έχουμε δηλαδή αφενός ε, τη μαζική παραγωγή και από την άλλη παραγωγή ε, μας πόρων συντηρών. Ε, θα πρέπει να υπάρξει χρήση της κόπριας που παράγει χιλιόμετρα. Είναι... Υπάρχει όμως η τεχνολογία. Είναι θέμα κόστους και θα πρέπει να υποστήριξουμε τους παραγωγούς και αυτή ακριβώ είναι η συζήτηση που γίνεται στην παρούσα φάση στη Γερμανία και περιέχει ακριβώ αυτή τη διάσταση του κόστου. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσέλερ. Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ε, όταν κοιτάμε, όταν επιτρέπουμε να υπάρχουν, ε, χρειάζεται να νοικιάσουμε ε, εκτάσεις για την κοπριά. Ένα λοιπόν ερώτημα είναι κατά πόσο θα έπρεπε να μειώσουμε την έκταση, το μέγεθος των... Ε, Πρέπει να γίνει μια διάκριση. Η Γεωργία έχει ως αποτέλεσμα την τέλημα ε, να χρησιμοποιεί λοιπάσματα για την ε, μεγαλύτερη απόδοση της γης και η κτηνοτροφία μπορεί να πάει. Οι χώρες που προσχώρησαν έπρεπε να φροντίσουν ε, κοντά σε μεγάλα ποτάμια να επεξεργάζονται τα λίματα. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον έγινε αυτό με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, αλλά το θέμα συχνά δεν είναι ή αν υπήρχαν δηλαδή. Και έτσι τα απόβλητα κατέληγαν ε, στα συστήματα υδρευσής ε, στο έδαφος, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν επαρκή ε, αγωγή. Το ίδιο έγινε και στον Βερολίνο το δεκαετία του Πολύ απλά λοιπόν αυτό που μας λείπει στο σημείο αυτό είναι μια γενική προσέγγιση. Παρευρεθήκαμε στο Κόνιξπερ Kaliningrad και τότε κάναμε και μια συμφωνία με την Ρωσία η οποία αναστάλησε μεταξύ περιλάμβανε πολλά χρήσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Καλινιγκράντ. Με μια αλυσίδα μέσα σε περιοχές να μην ε, περνάνε χωρίς καμία επεξεργασία στην ε, Βαλτική. Επίσης ε, με τη Ρωσία που είναι βασικός παράγοντας στην περιοχή και στο θέμα αυτό δεν έχουμε ουσιαστικές επαφές. Το 2009 ήμουν, αν θέλετε, πρότυπο αντιμετώπιση των μακροπεριφερειών. Τα προβλήματα της Βαλτικής ήταν και είναι γνωστά, ευτροφισμός, ε, μεγάλη επιβάρυνση με την κυκλοφορία των πλοίων, με τις, με την οποία είχαμε συμφωνία σύνδεση, ιατρική σχέση. Όλα αυτά βέβαια έγιναν ε, σε θεωρητικό επίπεδο. Θα τα έχουμε πετύχει μόνο αν όλοι όσοι είναι σε αυτή την μακροπεριφέρεια είχαν ε, δεσμευτεί για την εκπλήρωση των στόχων ε, που υπάρχουν στην πολιτική συνοχή και θα μπορούσαν να έχουν αφιερέσει πόρους. Αλλά δυστυχώ παρά τις ε, διασκέψεις, επιδιασκέψεων, δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Και αυτό φαίνεται. Η αλληλεία είναι το επόμενο θέμα και νομίζω ότι ότι θα έπρεπε να ληφθούν κοινά μέτρα. Όπως σας είπα, η μακροπεριφερειακή αυτή προσέγγιση έχει αποτέλεσμα μόνο αν δεσμευτούν όλοι οι συμμετέχοντες. Λέει πρόεδρος, δεδομένο και αυτονόητο. Ελπίζω να μην μας πάρει άλλα 10 χρόνια μέχρι ότου διαπιστώσουμε πάλι το ίδιο, να συνεχίσουμε Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση, την ευκαιρία να ακούσω τους προλαλήσαντες που έδωσαν τόσο χρήσιμα στοιχεία και σκέψεις. Νομίζω θα ακολουθήσω λίγο πολύ την ίδια γραμμή, στα έχω να πω και ξεκινώ με το υπόβαθρο. Εκπροσωπώ το πρόγραμμα EcoRegion για τη Βαλτική. Εργαζόμαστε εν γέννη σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ε, περιφερειακό συντονισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συγκεκριμένα για τη Βαλτική με τα γραφεία του WWF αλλά και ε, πέραν των χωρών της Βαλτικής και στο ε, Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας θέματα συνεργασίας και βιώσιμης διαχείρισης της Βαλτικής μας απασχολούν. Έγινε λόγος λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Βαλτικής, πόσο περίπλοκο είναι το πρόβλημα. Και κατέστησα σαφές ότι ο ευθροπισμός δεν οφείλεται μόνο στις συνθήκες στη θάλασσα αλλά και στη στερεά. Ο Κριστόφαλος θα ανέφερε νωρίτερα ότι είναι πολύ βραδύς ο κύκλος εναλλαγής των υδάτων και ανανέωσής τους. Άρα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι όλα αλληλένδετα. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει τεράστιες συνέπειες για τις χώρες σύλληψης είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από την ίδια την έκταση της Βαλτικής. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι τετραπλάσια η έκταση στη στεριά που επηρεάζει την Βαλτική και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε απα... απαντήσεις με μέτρα καθοριστικά κλείνοντας κάθε κενό που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Βαλτική. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω παραπάνω τον ευτροφισμό. Έχει καταστεί απόλυτο σαφές ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα και η γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο των αιτίων. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία με μια εικόνα πολύ συνηθισμένη. Έχουμε να κάνουμε με την παρουσία των φυκιών στην ε, Βαλτική μια ανοξική κατάσταση. Βακτήριο το οποίο τρώει το φύκι φτάνοντας μέχρι το βυθό. Και εδώ με τη φωτογραφία αυτή θέλω να σας εξηγήσω τι σημαίνει η, ε, ο ανοξικός βυθός. Φωτογραφία που μου έστειλε ένας ψαράς πέρσι, πρόκειται για γάδο, ένα από τα κύρια ήδη πολεύονται στη Βαλτική. Ο κοινό γάδο έχει συνήθω το ίδιο χρώμα. Το δεύτερο ίδιο που βλέπετε στο πλάι έχει το κανονικό χρώμα του ψαριού, στο μπούλχον. 40 μέτρα βάθος σε περιοχή ανοξική, δηλαδή με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο έχει αλλιευθεί το ψάρι αυτό και ενώ το, μόνο το πτερίγιο έχει το κανονικό χρώμα, το υπόλοιπο σώμα έχει αυτό το λευκό χρώμα με μόνο λίγο ε, μόβ στην μουσούδα που δείχνει πόσο ε, διαφορετικές είναι οι συνθήκες και πόσο επηρεάζουν τα ε, ψάρια. Εδώ έχουμε μια σειρά από κάρτες με ε, καταγραφή επιδόσεων, scorecards για να δείξουμε και το τι αποτελέσματα έχουν οι διάφορες δράσεις ε, με το σχέδιο δράσεως στη Βαλτική. Ξεκίνησαμε το 2007 εξετάζοντας την προόδο χώρα με βάση τις δεσμεύσεις αλλά και ευρύτερε δεσμεύσεις και διεθνείς για τον ε, χώρο των θαλασσών επί παραδείγματι, γενικά ευρύτερου, ευρύτερης κλίμακας δεσμεύσεις. Η Υπουργική απόφαση του Μαρτίου, πρόσφατα δηλαδή, έχει λάβει γνώση αυτών και ε, αυτές οι καρτέλες επιδόσεων μας οδηγούν πάντα στο συμπεράσμα ότι χρειάζεται ενίσχυση και της υλοποίηση των δεσμεύσεων, αλλά και πιο συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό δηλαδή που σας είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές πριν από μένα. Είναι πολύ σημαντικό όμως το να επισημαίνονται τα αισθήματα αυτά και από και οργανώσεις έξω από τον ε, χώρο άσκησης, χάραξης και άσκησης πολιτικής, αλλά και ευρύτερα για να γίνεται αντιληπτό το μέχρι που εκτείνεται το ζήτημα. Και πρέπει να εξηγήσουμε ότι μπορεί να έχουμε την πιο φιλόδοξη συμφωνία του κόσμου, αλλά εάν η υλοποίηση της δεν είναι εξίσου φιλόδοξη, αποτελέσματα δεν πρόκειται να φέρει. Μια πολύ σύντομη επισκόπηση λοιπόν σε σχέση με τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα δράσης για τη Βαλτική έχει τέσσερις τομείς ε, επιμέρους τομείς. Βλέπετε σε κόκκινο την αποτυχία στα συνολικά αποτελέσματα. Όλες οι περιοχές δηλαδή έχουν αποτύχει ως προς την υλοποίηση των, προ... τεσσάρων τομέων ε, στον σύνολό τους. Ε, μέχρι τώρα, γιατί η καταληκτική προθεσμία του 2021, όλες οι χώρες λοιπόν και οι περιοχές υπολείπονται των δεσμευσεών τους για τον ευτροφισμό. Βλέπετε βελτίωση σε κάποιες περιοχές και χώρες. Αναφέρθηκε και από την Επιτροπή ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην προσπάθεια αυτή η Δανία, αλλά και η Σουηδία και η Φινλανδία πάνε καλύτερα. Πάντω οι υπόλοιπε χώρε έχουν μάλλον αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορώ να σα δώσω αναλυτικά όλε τι διαφάνειες για τα διάφορα μέτρα αντιμετώπιση του ευθροφισμού αλλά στη θέση σα τα ε, έντυπα που έχω φέρει μαζί μου, σα ενδιαφέρει πλήρη έκθεση. Ε, έχουμε κάνει τρεις ε, ταξινομήσεις, τρεις κατηγορίες για τον ευτροφισμό, περιορισμό των ε, πηγών με μέτρα τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει οι χώρες πλην της Δανίας για τον περιορισμό των θρεπτικών ουσιών από αστικά λίματα μέσω από τις μονάδες καθαρισμού, για, τη, για, το γεωργικό, για τον περιορισμό των γεωργικών θρεπτικών ουσιών. Υπάρχουν κάποια μέτρα με αποτελέσματα όμω ανάμεκτα που απαιτούν περισσότερη δουλειά ακόμα. Κατευθυντήριε γραμμέ, προδιαγραφέ, η πρότυπα για την περιεκτικότητα τη θρεπτικής ουσία, οι παραδείγματα για τα λοιπάσματα, για τα φυσικά λοιπάσματα και περιορισμό τη ρήπανση από τη γεωργία. Εν ολίγη, επαναλαμβάνω αυτά που σα είπαν και οι προλαλήσαντες η γεωργία είναι ένας από τους κύριους τομείς τους οποίους πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, όπως άλλωστε και ο χώρος των αστικών λιμάτων, εκθέσεις του 2016 των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι αυτές τις οποίες έχουμε στηρίξει τα στοιχεία μας και δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε σχέση με τα όσα είπαν οι ε, προηγούμενοι ομιλητές νωρίτερα. Απλώς τα επικυρώνω και τα επιβεβαιώνω και εγώ εξεπλάγιν και κάτεπλάγιν που είναι τόσο κακά τα αποτελέσματα φαντάζομαι και εσείς και φαντάζομαι ότι θα μας ρωτήσετε γιατί όπως είπατε άλλωστε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 177 ήταν οι δράσεις για το πρόγραμμα δράσης της Βαλτικής εκ των οποίων οι 103 έχουν εκπνεύσει ήδη. Ε, από αυτές οι μισές 45 περίπου έχουν επιτύχει εν μέρη ή καθόλου τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή υπάρχουν άλλες τόσες που περιμένουμε να φέρουν αποτελέσματα. Αφενός με, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν εκούσες οι συμφωνίες, πολύ καλή σύμβαση, απαραίτητη, τη χρειαζόμαστε, μας έχει επιτρέψει να προχωρήσουμε πολύ, αλλά είναι μόνο σε εκούσια βάση. Και υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί από την άλλη που είναι πολύ ε, λιγότερο από απαιτητική, ενώ η Helcom όντας πιο απαιτητική είναι μόνο εκούσια. Ε, είναι μόνο σε θελοντική βάση. Και εδώ έχουμε και το πρόβλημα γιατί δίνονται διαφορετικές αποδόσεις αποτελεσμάτων από τη Helcom και αντίστοιχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράση, αλλά οι χώρες σε εθνικό επίπεδο δεν υλοποιούν αυτό το οποίο έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν. Και αυτό νομίζω το συζητήσαμε. Έρευνα πάλι. τεχνητά αλλά και φυσικά λοιπάσματα που δείχνουν ότι δεν ε, απορροφάται το υλικό το οποίο ε, ρίχνουμε πάνω στα φυτά το περισσότερο από το μισό περνάει στο έδαφος και μετά στα νερά, στα ύδατα και άρα πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια κυρίως στη στεριά και κυρίως σε σχέση με τη γεωργία. Υπάρχει επάρκεια σε θρεπτικές ε, ουσίες και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κυκλική οικονομία και για, την, ε, για το περιβάλλον νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και με μεγάλο κέρδος τόσο για το γεωργό ο οποίος δεν θα χρειάζεται πια να αγοράσει άλλο ε, αλλά και δίνοντας λύσεις πρωτοπόρες και οικολογικές για τη γεωργία μας. μιλήσαμε για περιβαλλοντικά προγράμματα και άλλα μέτρα που έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία, από τέλη τη δεκαετία του 90 και ήταν αποτελεσματικά γιατί στη τελευταία ανάλυση εξασφάλισαν καμιά ευαισθητοποίηση για το τι πρέπει να γίνει. Απλά πράγματα, αλλά όπω υπόθηκε και τα. Επίση έχουμε έναν διαγωνισμό. Ε, με τη βράβευση της, ε, του αγροκτήματος της χρονιάς της Βαλτικής ε, με τον Μάρκους Έρολα και τη Μινάσα Κέρολα που βραβεύτηκαν το 2015 γιατί αξιοποίησαν κάθε δυνατό μέσο ότι είναι δυνατό και μάλιστα το έκαναν μόνοι τους χωρίς να περιμένουν να τους ε, ε, το επιβάλλουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Και ξεπέρασαν αυτό το οποίο ήταν ε, οι υποχρεωτικές διατάξεις και υποχρεώσεις. Αυτή ε, το κατάφεραν λοιπόν, ολίγοι όμω είναι οι γεωργοί που κάνουν πραγματικά μέτρα ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η επάρκεια σε θρεπτικέ ουσίες. Καλά όλα αυτά που υπόθηκαν, αλλά νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές συμφωνούμε πως δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ευτροφισμού στη Βαλτική και η κοινή πολιτική νομίζω ότι είναι ένα από τα κύρια για τον διαπλαίσιο για τα αστικά λύματα. Ε, και, και άλλες αντίστοιχες, αλλά νομίζω το κύριο πρόβλημα, αυτό ίσως το οποίο πρέπει να καταδείξουμε και να ε, σταθούμε περισσότερο σε αυτό, είναι της κοινή ιερουργικής πολιτικής, γιατί αυτή είναι η πέτεια για το μεγαλύτερο μέρη του πλησμού της κοινή ιερουργικής πολιτικής. Στα δεξιά έχετε τις στήλες με πράσινο, τις πιο μεγάλες που είναι οι άμεσες ενισχύσεις και η τάση διατήρησης μέσα στην κοινή γεωργική πολιτική των άμεσων ενισχύσεων, υποστήριξη δηλαδή του εισοδήματο του γεωργού. Είναι το... Και νομίζω ότι η πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει μόλις κατατεθεί, ίσως δώσει κάποιε απαντήσεις για το πρόβλημα αυτό. Για εμά, για την WWF, είναι πολύ σημαντικό οι ενισχύσεις που θα φτάνουν στο Γεωργό οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Τα μέτρα περνούν μέσα από τη γεωργική πολιτική σε όρους εθελοντικούς και μέσα από το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. Ωστόσο σε αυτό, όπως έχει διατυπωθεί τώρα, μόνο 30% των ε, ποσών πρέπει υποχρεωτικά να αξιοπορούν συνεργατικά, ε, να δώσουν συνδυασμένες, να δώσουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια έκθεση έρευνας από το κέντρο AgriFood, οικονομικό κέντρο AgriFood της Σουηδίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με μικρότερο περιβάλλον με μικρότερο προπολογισμό. Και όντω θα είναι μικρότερο ο προπολογισμό, αυτό βλέπουμε ήδη. Χρειάζονται όμω αλλαγές σε σχέση με την ε, κατάρτιση των άμεσων ενισχύσεων. Πρέπει να βρεθούν δηλαδή διαφορετικοί τρόποι χρήσεως των κονδυλίων αυτών. Εδώ στην έκθεση, από την έκθεση αυτή, την AgriFood, έχω αντλήσει κάποιες ε, ενίσχυση παραδείγματι σε ζώνες που έχουν υψηλή ε, γεωργική αξία ή μάλλον φυσική αξία ή επίσης μέτρα, ένα θέμα πιο σχετικό με το δικό μας ε, ζήτημα σήμερα, για την αποτροπή του ευτροφισμού που να βοηθήσουν στον περιορισμό. Αλλά γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κίνητρο προς το Γεωργό να περιορίσει τη χρήση των φυσικών λιπασμάτων που χρησιμοποιεί. Και άρα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για περιορισμό των ε, αιτίων του ευτροφισμού. Για να κλείσω λοιπόν ε, εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην περιοχή. Χρειάζεται να υλοποιηθούν μηχανισμοί για την αποτροπή εξελίξεων που ε, είναι στρεβλές. Πρέπει δηλαδή στοχευμένα να δίνουμε τα χρήματα, ε, να διατίθεται τα χρήματα εκεί που πραγματικά χρειάζονται και με, τους, με το κατάλληλο αποτελέσμα. Χρειάζεται μια ποιότητα των έργων της ε, ΚΑΠ ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι και αυτό ήταν το τέλος της παρουσίασης μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σήμερα. Ασχοληθήκαμε με την ε, ΚΑΠ και θα είχαμε διάφορες προτάσεις να κάνουμε για τη βελτίωση της ΚΑΠ. Γι' αυτό λοιπόν τα σημειώνουμε με χαρά την ε, Interreg ε, για την ε, Νότια Βαλτική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Εκπροσωπώ το πρόγραμμα Interreg, την Κοινοτική Πρωτοβουλία για τις Παραμεθόριες Περιοχές στη Νότια Βαλτική. Θα σας μιλήσω όμως παρεμπιπτόντως και για διάφορα προγράμματα Interreg. Η παρουσία μου έχει στοιχεία και από άλλα προγράμματα Interreg. αλλά δεν αντικατοπτρίζει πάντα την επίσημη θέση. Οπότε λάβετε το αυτό υπόψη. Θα ήθελα πρώτα να σας εξηγήσω τι εστί interreg, πώς λειτουργεί γενικώ και πώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του ευτροφισμού. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα σχεδίων του interreg και μετά θα σας παρουσιάσω και κάποια προβλήματα ή τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Τι είναι Ιντερεκ το, τα προγράμματα Interreg στόχο έχουν την επίλυση κοινών ή παρόμοιων προβλημάτων παραμεθόριων περιοχών σε περίπτωση που τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να επιληθούν σε μια μεμονωμένη χώρα. Στόχος των προγραμμάτων Interreg είναι να αναπτύξουν λύσεις, να μεταφέρουν γνώση και να διαδώσουν τις γνώσεις και τις νέες λύσεις. Καταρχήν, το πρόγραμμα Interreg δεν χρηματοδοτεί βασική έρευνα, οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιο στοιχείο, εφαρμογής η πιλωτική δοκιμασία, πειραματική δοκιμασία νέων τεχνολογικών λύσεων, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε τεράστιες επενδύσεις ε, ούτε σε υποδομές ε, δυνάμει των προγραμμάτων Interreg. Και ε, ίσως και λόγω αυτού του στοιχείου δεν είναι άμεσα τα αποτελέσματα των σχεδίων Interreg. Τα προγράμματα του Interreg ε, διακρίνονται σε διακρατικά και σε διαμεθοριακά, διασυνοριακά. Τα διακρατικά ε, περιλαμβάνουν ολόκληρες χώρες, ενώ τα διασυνοριακά συνήθως περιλαμβάνουν μόνο τις παραμεθόριες περιοχές. Είναι συμπληρωματικά τα διακρατικά και τα διασυνοριακά σχέδια. Συνήθως τα διακρατικά ε, γίνονται μεταξύ Υπουργείων και Περιφερειακών Αρχών, ενώ τα διασυνοριακά προγράμματα πολύ συχνά στοχεύουν σε τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το σημαντικό πάντως είναι ότι τα προγράμματα Interreg καλύπτουν διάφορα θέματα. Ανάπτυξη επιχειρήσεων, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παιδεία, μεταφορές, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα. Η συνήθις ε, δομή των προγραμμάτων Interreg ε, προβλέπει στρατηγικές αποφάσεις να λαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης που απαρτίζεται από εκπροσώπους των περιφερειών. Γιατί αυτοί λαμβάνουν την απόφαση για το τι θα χρηματοδοτηθεί σε δεδομένο πρόγραμμα. Στην περιοχή της Βαλτικής, στην περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας, έχουμε πάνω από 12 προγράμματα Interreg. Τα περισσότερα τα βλέπετε εδώ στο χάρτη. Είναι 7 θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία και 5 χερσαία διασυνοριακή συνεργασία. Με σαφή εστίαση σε θέματα ευτροφισμού μόνο σε τρία από τα προγράμματα αυτά. Το μεγαλύτερο καλύπτει σχεδόν μια ολόκληρη περιφέρεια που αναφέρεται, βλέπετε και στη διαφάνεια, αφορά τη Βαλτική ε, το μπλε είναι η Νότια Βαλτική και το πράσινο είναι το διασυνοριακό πρόγραμμα της Κεντρικής Βαλτικής. Εγώ εκπροσωπώ το πρόγραμμα της Νότιου Βαλτικής. Περίπου 14 δισεκατομμύρια, όπως ακούσαμε, αφιερώθηκαν στο, στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 για τα θέματα της, ε, του ευτροφισμού, πάνω από 14 και το Interreg είναι ένα μικρό κλάσμα αυτής της χρηματοδότησης. Πάντως σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ότι τα τρία προγράμματα που στόχο έχουν την καταπολέμηση του ευτροφισμού από το 2007 έχουν αφιερώσει από ένα τέταρτο μέχρι το μισό προϋπολογισμό τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Ένα τέταρτο με το μισό προπολογισμό αφιερώθηκε στην καταπολέμηση του ευτροφισμού και μέσα σε μία δεκαετία 43 σχέδια 80 εκατομμυρίων αξίες, ε, εφαρμόστηκαν από αυτά τα τρία προγράμματα Interreg. Τώρα, τι γίνεται από το σύνολο του προγράμματων των Interreg στη Βαλτική. Τα τρία αυτά προγράμματα Interreg παρέχουν το 90% της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του ευτροφισμού και πάρει ένα μικρό, κλάσμα του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού της εθνικής χρηματοδότησης, αλλά για τις διασυνοριακές ε, ε, μεθόδους συνεργασίας ε, είναι αρκετά σημαντικό αυτό το μερίδιο. Ο ρόλος των προγραμμάτων αυτών είναι να δοκιμάσουν νέες λύσεις ή να μεταφέρουν ή να εφαρμόσουν νέες λύσεις σε τοπικές ε, περιοχές και διασυνοριακά. Τώρα ως προς τα σχέδια, κάποια παραδείγματα σχεδίων. Τα περισσότερα σχέδια επικεντρώνονται σε δύο τινά. Είτε στην αποτροπή της ε, απόρριψης ε, θερεπτικών ουσιών, είτε στα υπόγεια ύδατα, είτε στη θάλασσα, είτε στην απομάκρυση, αφαίρεση θερεπτικών ουσιών που ήδη έχουν κατακαθίσει στη θάλασσα σε κάποιες μολυσμένες περιοχές της Βαλτικής. Εδώ σε αυτή την φωτογραφία βλέπετε ένα παράδειγμα του σχεδίου που αφορά στα διαχειριστές σταθμών επεξεργασίας αστικών λιμάτων που ασχολούνται κυρίως με την απόρριψη φαρμακευτικών ουσιών μέσω των λιμάτων προς τη θάλασσα. Στόχος λοιπόν είναι να γίνει ένας απολογισμός των ε, τεχνολογιών επεξεργασίας για να δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές από άποψη κόστους. Και μια και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βαλτική που αναφέρθηκε, αυτό είναι ένα εμβληματικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την μακροπεριφέρεια της Βαλτικής. Το επόμενο θα το παρακάμψω. Εδώ έχουμε τις ζωντανές λιμνοθάλασσες, το σχέδιο Live Lagoons, που στόχο έχει την αφαίρεση θρεπτικών ουσιών από τη θάλασσα. Έχει μόνο τοπικό αντίκτυπο αυτό το σχέδιο, αλλά ο στόχος του είναι να δοκιμάσει αποτελεσματικά ψηκό στους μέτρα για την αφαίρεση θρεπτικών ουσιών. Με την εγκατάσταση, για παράδειγμα, πλωτών νήσων ε, υγροτόπων που απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες από το νερό. Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα μιας πλατφόρμας για τη διασύνδεση πηγών για την αφαίρεση θρεπτικών ουσιών με ε, εκούσια βάση είναι παρόμοιο με τις αντισταθμίσεις ε, της εμπορίας εκπομπών μεταξύ των ρηπενόντων και των πηγών ε, των τεχνολογιών ε, απομάκρυνση των θρεπτικών ουσιών. Και πρόκειται για ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από το Interreg ε, τη Κεντρική Βλακτική και είναι εμβληματική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την μακροπεριφέρεια τη Βαλτική. Επόμενο θέμα είναι ένα παράδειγμα σχεδίου ενός project που θέλει να αντιμετωπίσει τις διάχυτες πηγές ρήπανσης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αυτό, αλλά είναι ευρύ το φάσμα αυτού του project. Είχαμε 170 πρότυπες γεωργίας εκμεταλλεύσεις σε 7 χώρες της Βαλτικής και ε, δοκίμασαν και παρουσίασαν τα πιο φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα για τη μείωση αυτών των απολύων θρεπτικών ουσιών. Και μάλιστα τα αποτελέσματα της, ε, του πειράματος αυτού διαδόθηκαν σε περίπου 2.500 γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τον τρόπο μείωσης των απολειών από θρεπτικές ουσίες. Ένα από τα προβλήματα και πιθανή βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί αφορά το νομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι ο Μεγαλύτερο πονοκέφαλο της κοινότητα του Ιντερεκ είναι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που έχουμε καταρχήν ε, μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμοστεί με ένα σχέδιο με κρατική ενίσχυση και αποτρέπει μερικούς ενδιαφερόμενους από την εμπλοκή στο πρόγραμμα, στο σχέδιο. Γιατί οι διατυπώσεις, οι διοικητικές διατυπώσεις για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης είναι δυσάρεστες. Και ας σκεφτούμε και την κλίμακα, τότε δεν αξίζει όλη η προσπάθεια. Δεν αξίζει τον κόπο. Και αν δεν υπήρχαν κρατικέ ενισχύσει, θα είχαμε πολύ περισσότερα προγράμματα Ιντερνετ και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τι πειραματικές δοκιμές και τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στα προγράμματα αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι ότι έχουμε πολύ άριθμα προγράμματα Interreg που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον ευτροφισμό και η διαπρογραμματική συνεργασία δεν έχει φτάσει σε καλό επίπεδο ακόμη. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία αυτής της συνεργασίας μεταξύ των προγραμμάτων και να συνδυάσουμε κάποια mainstream κονδύλια και διεθνή κονδύλια, ώστε να τα συμπεριλάβουμε στο νομικό πλαίσιο. Βέβαια το ότι έχουμε πολλά προγράμματα δεν είναι κατά ανάγκη κακό, γιατί έτσι μπορούν ε, και οι περιφέρειες να εμπλέκονται περισσότερο και να κάνουν κτήμα τους ε, τα προγράμματα συμμετέχοντας στη, στη λήψη των αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τα πλαίσια πολιτικής και αυτό το θέμα τη σχέση των προγραμμάτων με το πλαίσιο πολιτικής θα μπορούσε να βελτιωθεί. Καλύτερη συμπερίληψή τους στα πλαίσια, τα νομικά πλαίσια. Αν και το προσωπική μου γνώμη είναι ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι και πολύ άσχημα, γιατί πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούμε τη χάνουν τη υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Βαλτική Θάλασσα. Υπάρχει συνεργασία με άλλες πολιτικές. Τώρα το θέμα της απλούστευσης, τη της απλούστευσης των κανόνων χρηματοδότησης. Ε, συνεχίζεται η συζήτηση για το θέμα αυτό, οπότε δεν θα εντρυφήσω ιδιαίτερος. Απλούστεροι κανόνες για την ε, ε, εισπράξη των κονδυλίων. Η καλύτερη προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Σε ό,τι αφορά τις δυνητικές βελτιώσεις του προγράμματος, θα έλεγα ότι το μείζον που αφορούν κυρίως την διάδοση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και του αντικτύπου τους. Γιατί συνήθως όταν ε, εξαντληθούν τα κονδύλια υπάρχει μια διαφορία για τα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν τα προγράμματα να κεφαλαιοποιήσουν περισσότερο, να το βελτιώσουμε. Καλύτερη διάδοση και καλύτερη κεφαλαιοποίηση, καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, χάρη στην ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Παράδειγμα, μια πρωτοβουλία που εφαρμόσαμε στη Βαλτική με τίτλο «Πλατφόρμες προγραμμάτων» άλλα κονδύλια και που μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικά κονδύλια για να εφαρμόσουν συνεργασία μεταξύ τους. Έτσι αξιοποιούνται καλύτερα οι, οι βέλτιστες πρακτικές και δοκιμάζονται σε διαφορετικούς. Ε, η πλατφόρμα των σχεδίων έχει ξεκινήσει ήδη μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη Βαλτική θάλασσα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η απόφαση θα ληφθεί τον Ιούνιο του 2018 για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά ευχαριστώ. Για το τρίτο τμήμα της ακρόασης δεν έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις να κάνω. Μία μισή ερώτηση, μισή σχόλια, αν μου επιτρέπετε, προς την κυρία Γιατί παρουσία Τα σημειώνουμε τα σημεία αυτά και φυσικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Περιμέναμε μια δραματική παρέμβαση στον τρόπο διαμόρφωσης του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων. Μήνυμα που έστελνε επί σειρά ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο για όλα αυτά. Προσεκτικά αυτά που προτείνεται είναι σαφέστατη, όμω δεν έχω άλλε ερωτήσει να κάνω. Ίσως κάποια, κάποια βουλευτέ. Οι μη κοινότητε θα ήθελαν να συμμετάσχουν πιο πολύ, αν το μπορούσαν. Τι προγράμματα έχετε υπόψη σα ό,τι αφορά Κοιτώντα την κλίμακα ενό έργου. Συνήθω μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Γιατί ε, οι κρατικές ενισχύσεις ε, αποτρέπουν οποιαδήποτε ανάμειξη. Γιατί η γραφειοκρατία που συνδέεται με τους κανόνες για την κριτική ενίσχυση είναι πραγματικά πολύ υψηλή και δεν μπορεί να την διαχειριστεί μια μικρότερη οργάνωση που πολύ απλά δεν θέλει να συμμετάσχει στα προγράμματα. Δεν ξέρω αν σωστά κατάλαβα την ερώτησή σας. λέτε για την κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για τη μεγάλη, ε, η μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγόντων. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι οριακέ τιμέ θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλέ. Στην ευρυζωνικότητα το έχω πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό. Ούτε οι δήμοι το τολμούν, γιατί έχουν κάποιο άλλο το ποσό. Δεν θέλω να κάνω λανθασμένες συνδέσεις, απλά θα θέλω να μου πείτε τι ακριβώς εννοείται, γι' αυτό και ζήτησα να το ευκρινίσετε. Και ο συναδελφός Τσέλερ έχει να κάνει μια ερώτηση για το θέμα αυτό. Όταν η ίδρυυση και η επεξεργασία των λιμάτων σε μια περιφερεια είναι στα χέρια των Δήμων, αλλά οι επενδύσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρέ κομμοπόλεις, για παράδειγμα, τα συστήματα λοιπόν και ε, με τους κανόνες για τον οργανισμό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί διαρκώς στην περιφερειακή πολιτική, κατά πόσον οι μηχανισμοί υποστηρίξουν. Δεν φτάνει να υπάρχουν μεγάλα προγράμματα για την ε, επεξεργασία υδάτων σε κάποιες χώρες και να μην υπάρχει το κρατικό ή δημοτικό για την αποχέτευση, το οποίο θα συνδεθεί στην, στην εγκατάσταση εργασία λιμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς ε, να διοχετευτούν τα λύματα προς τις καταστάσεις. Παρατήρηση σε σχέση με το πόσο περίπλοκο είναι όπως διαπιστώνουμε το σύστημα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς ε, υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των ε, εισρεών των ποσών εισρεών στη γεωργική πολιτική δηλαδή και της ποιότητας του περίπτωση χρόνια και επίσης αυτό που παραμελήσαμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχει και η φύση τους κανόνες της. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα με τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν σήμερα. Ε, μπορώ να σας δώσω όμως και ένα άλλο παράδειγμα, Πρόεδρε. Ο Δήμος μου, ε, γεωργική άρτευση κτλ. Και, και μάλιστα αντί για μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, στην περιοχή γύρω από την λίμνη αυτή, φυτεύτηκε καλαμπόκι. Ε, αντιμετωπίσει την ύλη που ξεχύλισε και δεν μπορούσαν να επιδότηση απευθείας, ε, ανακαλύφθηκε ότι ήταν μολυσμένη αυτή η ύλη και έπρεπε να αφαιρεθεί και να αποτεφρωθεί. Αυτό λοιπόν για να δείξουμε ότι σε μια θάλασσα φαίνεται να ψοφούν σε μια συγκεκριμένη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι δεν σουφούν και αλλού τα ψάρια. Ναι, αυτό που θέλουμε να πούμε με την ε, διαφάνεια αυτή ήταν ότι οι εργασίες ή τα έργα στο καταρχήν δεν είναι αρκετού μεγέθους ώστε να επηρεάσουν τις συνθήκες της αγοράς. και από τα όσα έχω δει στις διάφορες συνεδριάσεις νομίζω μπορώ να επισημάνω ότι η κλίμακα δεν είναι τέτοια που να κινδυνεύει να καταστρέψει συνθήκες της αγοράς. Αυτό κλειστή να απαλλαγεί το ίντερνετ από τους όρους για τις κρατικές ενισχύσεις, για τους κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις. Καλώς, ολοκληρώσαμε το πρόβλημα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για μια φορά να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας. Εγώ καταγράφω τα εξή από τη σημερινή συζήτηση. Χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγέ να από τον κύριο Χόμπολτ. Σε Τα πάντα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πιο αυστηρή νομοθεσία. Σε σχέση με το πολιτεύσιμο νομικό πλαίσιο και την κυριαρχική πολιτική, πρέπει να κοιτάξουμε και τις, τους όρους ερεσιμότητας. Επιλέγουμε να ε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Γιατί βέβαια είναι σημαντική η πόρη που παίρνουν τα κράτη αυτά. χρησιμοποιηθούν μέτρα αποτελεσματικά. Και πρέπει βέβαια και εμείς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε βέβαια σε το χρόνο. Σας υπόσχομαι ότι θα διατηρήσουμε την επαφή. Θα κάνουμε... Βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να υπενθυμίσει το θέμα των επιζήμινων ουσιών τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα χρήσιμο των έργων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ναι, ευχαριστώ. Εκ μέρους της ε, κυρίας Λερόγεβε που είναι η Σκιώδης έχω να κάνω μια δήλωση. Κύριε Πρόεδρε, με εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, με το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ θετική έκθεση. Με ικανοποίηση παρακολουθούμε θετικά αποτελέσματα. Εν γένει ως μέλος ε, της Επιτροπής Επασχόλησης με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ικανοποίηση την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών, ιδιαίτερα από την στιγμή που έχει καταστεί μέλος της Επιτροπής ε, ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προτείνει και επιμένει ότι πρέπει να ε, μαθαίνουμε από τα σφάλματά μας και να τα διορθώνουμε και επιπλέον πρέπει να στηριζόμαστε και στα διδάγματα του παρελθόντος. Συστάσεις για τα κράτη-μέλη βέβαια, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτές. Επίσης, συνάδελφος ε, ελπίζει ότι θα εστιάσουμε καλύτερα την προσοχή μας σε αποτελέσματα και διαδικασίες επιλογής με την ε, επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων μόνο όταν αυτά έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα να παρουσιάσουν με βάση και την ειδική αυτή έκθεση. Θέλει να υπογραμμίσει τη σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ως ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας από τα 40 έργα 13 δεν, δεν θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 18 θα είχαν εκτελεστεί αλλά με περιορισμένη κλίμακα και χρονοδιάγραμμα και ορισμένα ε, ακόμη και χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί. Αυτό ε, πρέπει να καθοδηγήσει και την εστίαση των στόχων μας για το πολιτική πολιτές στο πλαίσιο και προσβλέπει στη συνεργασία με τον Ιστό. Πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κυρίε και κύριοι βουλευτέ εκ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, καλωσορίζουμε την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι ε, παραγωγικέ επενδύσει για τι επιχειρήσει, η οποία έκθεση συμβάλλει στην υποστήριξη των δικών μα προσπαθειών ε, για την επίτευξη μια νοοτροπίας αξιολόγηση με βάση τις επιδόσεις. Εμείς ε, εδώ αναγνωρίζετε ότι το ε, κανονιστικό πλαίσιο για την βιωσιμότητα των παραγωγικών επενδύσεων έχει βελτιωθεί με την, μέσα από την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι παρόλα αυτά χρειάζονται παραπάνω δράσεις για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και στην τρέχουσα ε, προγραμματική περίοδο που θα παρουσιάσει κάποιε καθυστερήσει, αλλά και για να επιτυχηθούν ακόμα προ διαδικασίε στο προσχέσει πολιτή οικονομικό πλαίσιο και το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε υποστήριζε την βιωσιμότητα και τη διάρκεια τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με την εγκαθίδρυση μια κοινή στρατηγική προσέγγιση ε, και προγραμματισμού και μέτρων συνοδευτικών, ειδικότερα ωστόσο. Έχουμε εγκαθιδρύσει μέτρα όπως την εκ των προτέρων αξιολόγηση για την ανάλυση κόστου αποτελέσματος για τα μεγαλύτερα περισσότερο χαρακτήρα έργα, συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης εποπτείας για την παρακολούθηση και εποπτεία της προόδου και ιδιαίτερα σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων, νέες προϋποθέσεις για τα κράτη-μέλη που απαιτούν την ε, διεξαγωγή τουλάχιστον μίας ε, αξιολόγηση των άξιων προτεραιότητας και προσέγγιση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς μια συστηματική ε, ανάλυση εκ των υστέρων, αξιολόγηση εκ των υστέρων και βεβαίως σε σχέση με την επιμερισμένη διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι με την αρχή αυτή πρέπει και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν την ε, διάρκεια των αποτελεσμάτων με επιλογή προσεκτική, με βάση κριτήρια, με βάση το, την νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται. Και για να πω δύο λόγια για την έκθεση και τη σύσταση. Και Τα πορίσματα του Ευρωλεκτικού Συνεδρίου δείχνουν ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι πολιτικές προϋποθέσεις σε κάθε έργο που ελέγχθηκε, έχουν ε, γενικά αποδώσει τους αναμενόμενους στόχους και μάλιστα ε, και μέσα στις ε, προθεσμίες που είχαν προσδιοριστεί. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα δεν διατηρήθηκαν τα αποτελέσματα σε ορισμένε περιπτώσει, και αυτό οφείλεται σε, μεγάλο, σε ένα βαθμό στην έμφαση που θα έπρεπε περισσότερο να είχε δοθεί από τη διαχείριση του προγράμματο στην ε, αηφορία, στη διάρκεια και επίση εξωγενείς σε ορισμένες παρα... περιπτώσεις ε, παράγοντες όπως οι οικονομικές συνθήκες ή συνθήκες αγοράς που είχαν αρνητική επίπτωση στην διάρκεια ορισμένων προγραμμάτων. Έχουμε πέντε, καρονες, πέντε συστάσεις ε, προς τα κράτη-μέλη, τρεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται και τις τρεις συστάσεις που την αφορούν σε σχέση με την προαγωγή του, της, απόδοσης και, ε, της ε, διάρκειας της απόδοσης και, της αποτελεσμα, και των αποτελεσματών με, την εκ των υστέρων αξιολόγηση μετά το πέρας της περίοδου αλλά και την εισαγωγή διορθωτικών μέτρων Δεσμεύομαι λοιπόν εδώ πως ιδιαίτερη προσοχή πρόκειται να δώσουμε στο ζήτημα της ε, ικανοποίησης του όρου της διάρκειας έναντι των άμεσων αποτελεσμάτων τα κράτη-μέλη. Και ιδιαίτερα στα προγράμματα που ισχύουν για την περίοδο μετά το 2020 πρόκειται να ενισχύσουμε την ε, ε, ε, ανάλυση της διάρκειας, ε, της ανθεκτικότητας στην ε, εκ των υστέρων ανάλυση. Βέβαια αυτό πάντα θα εξαρτάται και από τον τύπο, τη διάρκεια και τον τύπο αξιολόγηση και το χρονικό σημείο της αξιολόγηση. Και επίσης μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το άρθρο 71 θα τηρείται και τηρείται ήδη με αυστηρότητα, δηλαδή θα κάνει καθαρές διορθώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την διάρκεια. Ευχαριστώ. Κύριε Μπάλκο, θέλετε να πάρετε το λόγο πάλι. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα των όσων ε, κοιτάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και πώς μπορείτε εσείς ως νομοθετικό σώμα να βελτιώσετε τη δαπάνη των ε, πόρων αυτών το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει επιφέρει βελτιώσεις. Για την περίοδο 2013 θα είσαστε βασικό ε, φορέας για την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Με την έκθεση λοιπόν αυτή μπορείτε να έχετε ένα εργαλείο στη διάθεσή σας για να βελτιώσετε την κατάσταση την επόμενη φορά. Εμείς ε, ασφαλώς ε, είμαστε στην διάθεσή σας να παρουσιάσουμε εκ νέου την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μόνο εμάς. Εξίσου θεωρώ ότι απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσά. Ευχαριστώ. Το κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι από όλα όσα ακούσαμε η... Ακριβώς αυτό το στόχο θα επιδιωκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώσαμε και το 13 της ημερήσης διάταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσουμε στο 14 η ημερήσης διάταξη για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η κυρία Κάντεμπαχ είναι η συγγήτριά μας και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φιγκρέδο από το ανεκτικό Συνέδριο. Thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, πριν κάνω τη σύντομη παρουσίαση, να τονίσω ότι επανερχόμαστε στο θέμα της ΚΑΠ, της κοινής γεωρικής πολιτικής και τονίζουμε κάποια θέματα που αφορούν την απλούστευση και την καλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα. Αυτή είναι η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαμε σε πολλά κράτη-μέλη για τις νέες απλουστευμένες επιλογές κόστους. Όπως ξέρετε, οι παραδοσιακές λύσεις για την χρηματοοικονομική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης είναι η επιστροφή των δαπανών που έγιναν και επανειλημμένω το Ανακτικό Συνέδριο στο παρελθόν έχει πει ότι τέτοιου είδου ε, παραδοσιακέ λύσει ε, είναι επιρρεπεί στα σφάλματα. Γι' αυτό και ελπίζουμε και πιστεύουμε ακράδαντα ότι καλές λύσεις μπορούν να προέλθουν ή τυποποιημένε κλίμακες μοναδιαίου κόστου. Και ε, εξυπηρετούν καλύτερα του τελικούς δικαιούχου και συνάδελφους. Αυτά τα μέτρα και των νέων λύσεων για τις πληρωμές, για τις ενισχύσεις ή της χρηματοπιστωτικής ε, ε, στήριξη. οι επιλογές απλουστευμένου κόστους μετά την διεκπαιρέωση του ελέγχου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι, ε, επιλογές απλουστευμένου κόστους ε, αποτελέσματα, με εγκάρση αποτελέσματα. Τώρα δούμε τη χρήση αυτών των ε, επιλογών απλουστευμένου κόστους και πόσο συνάδουν με την ΑΚ και επίσης έχουν απλουστεύσει τις διοικητικές διατυπώσεις, γιατί οι διοικητικές αρχές κατά τη, κατά τη διενέργεια των διοικητικών και εκεί βρήκαμε καλά παραδείγματα μεθοδολογίας και υπολογισμών, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ε, τα, δεν είχαμε αρκετά δεδομένα. Ή δεν... Πάντως ένα θέμα που θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή είναι ότι βρήκα αργές απλουστευμένου κόστους για να ε, γενικευθεί η χρήση τους από τα κράτη-μέλη και τις ε, διοικήσεις. Πάντως, δύσκολη τη χρήση των ΕΑΚ, αλλά μπορούν παρόλα αυτά να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων αυτές οι επιλογές απλουστευμένου κόστους. Τελέσματα με καλύτερη στόχευση τα αποτελέσματα συνδέθηκαν με ε, την, την έκβαση αλλά όχι τα αποτελέσματα. Οπότε, η πρώτη μας σύσταση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, ενημερώσει, να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ΕΑΚ, να ε, διευκρινίσει τις ε, αρχές πιστοποίησης και να περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των ΕΑΚ στα αισθήματα ελέγχου και τέλος, τρίτη και τελευταία σύσταση, συστήνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την κατάλληλη χρήση των ΕΑΚ, των επιλογών απλουστευμένου κόστους, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει την πιθανότητα περαιτέρω ανάπτυξης ε, ε, γιατί απλοποιούν. Είναι πιο απλό και για την, ε, τις αρμόδιες αρχές, αλλά και για τους τελικούς δικαιούχους, φυσικά. Και αυτό συνδέεται με τη δεύτερη ερώτηση την οποία κάνατε. Εδώ σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των απλοποιημένων εκδοχών. Γιατί θα χρειαστούν, θα πρέπει να αναπτύξουν ιδιαίτερη μεθοδολογία για να δημιουργήσουν αυτές τις αναλλακτικέ λύσεις και να πούν ποιου μηχανισμού συγκεκριμένα κάνουμε του ελέγχους μας. Είναι το εξή. Παρά το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η επιπρόσθετη δυσκολία στην αρχή για τι υπηρεσίε, σε τελική ανάλυση Δεδομένων όλων των διαδικασιών, αυτές οι λύσεις τελικά αποδεικνύονται πιο απλές και για τις υπηρεσίες. Είναι πιο απλές και πρέπει να αναπτυχθούν, να, πρέπει να υποστηριχθούν στην αναπτύξη της υπέθρου, Σύμφωνα και με τα παραδείγματα που έχουμε δει και σε άλλες πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η πολιτική συνοχή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Η δεύτερη σύσταση τώρα είναι κεντρικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των νέων των εναλλακτικών Το θέμα της μεθοδολογίας είναι εγγενές. Γιατί οι μεθοδολογίες υποστηρίζουν την ορθότητα της α, οικονομικής ανίσχυσης και άρα θα πρέπει να είναι ορθές και εύρωστες. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σαφές που είναι πίσω από τις λύσεις αυτές είναι καλά σχεδιασμένες. Δεν ξέρω αν απάντησα με τον τρόπο αυτό στην ερώτησή σας, γι' αυτό λοιπόν και προβήκαμε στην σύσταση αυτή. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι κάποια, να υπάρχει κάποια παρανόηση. Εγώ δεν ανησύχησα. Εδώ συμφωνούμε, λέει η Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση. Αγκρή. Μιλούσε. Πέρασε, παρακαλώ.